Buenas tardes. Vamos tomando asiento. Καλησπέρα. Καθίστε. Ας ξεκινήσουμε με την ακρόαση αυτή. Για την αλία στα βαθιά νερά. Καταρχά να σα ευχαριστήσω όλου για την παρουσία σα εδώ, ιδίω ε, του εισηγητέ σε ένα θέμα που είναι γεγονός ότι είναι σημαντικό, ενδιαφέρον και ιδίως περιλαμβάνει πολλά θέματα για συζήτηση. Το ότι καταφέραμε νομίζω να συναντηθούμε ε, εμπειρογνώμενες από διάφορους κλάδους που θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε κάτι καλύτερα την πρώτη της Επιτροπής θα είναι καθοριστική σημασία και νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο γίνεται την σημερινή συνάντηση είναι γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής ε, είναι αμφιλεγόμενη. Κάποιοι είναι πολύ υπέρ του να απαγορεύονται ε, τα, τα απλάδια ή τα απλάδια βυθού, αλλά και είναι άλλοι που είναι αντίθετοι. Πάντως είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή εικόνα. Μέχρι τις 6.25 χρόνο έχουμε. Η προσέγγιση που ακολουθούμε, σύμφωνα με τους συντονιστές, και σας το λέω να το ξέρετε κι εσείς, είναι πρώτον, βεβαίως θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ασένη για μια σύντομη εισήγηση. Κατόπιν έχουμε τέσσερα χωριστά πάνελ, με δύο παρεμβάσεις σε κάθε πάνελ πέραν των δύο ατόμων ανά πάνελ, που θα είναι οι εισηγητές, έχουμε και ένα καινούριο στοιχείο. Έχουμε παρουσία και παρέμβαση τεσσάρων ακόμα συν εισηγητών, παρεμβενόντων, που θα λάβουν το λόγο για το ίδιο θέμα. Ανάλογα με το πώς πάει η κατάσταση, ή στο τέλος του δεύτερου ή στο τέλος του τέταρτου, ε, θα δούμε. Μετά από κάθε πάνελ θα υπάρχει και μια σειρά ερωτήσεων και παρεμβάσεων των βουλευτών που θα μπορούν να θέσουν ερωτήσεις. Στο τέλος του του πάνελ, στο τέλος δηλαδή της ε, αν έχει χρόνο, αν έχουμε χρόνο που το ελπίζω και αν περιοριστούμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και στο χρόνο που μας έχει δοθεί θα υπάρξει ένας ανοιχτός κύκλος παρεμβάσεων όλων όσοι θέλουν να μιλήσουν, είτε βουλευτές, είτε όχι. Πάντα βέβαια εφόσον υπάρχει επαρκής χρόνος. Στο τέλος. Νομίζω ότι είναι σαφές ε, το πλαίσιο. Αν εφετέρου, επαναλαμβάνοντας ευχαριστίες ε, προς όλους, είναι το λόγο στον κύριο Ασένη εισηγητή για το θέμα. Κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε εδώ ε, για να συζητήσουμε ένα χαρακτηριστικό, ένα σημαντικό θέμα της αλίας. Η αλία των βαθιών υδάτων κατ' ουσίαν ε, αποδεικνύει το τι συμβαίνει γενικότερα στην Αλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, η αλία γίνεται άκρητα με αποτέλεσμα ορισμένα θέματα να εξαντλούνται και συμβαίνει και το αντίθετο. Έτσι λοιπόν ε, ε, όταν βλέπουμε βενθοπελαγικά είδη ε, ψαριών τσαντλούνται τα αποθέματα τους ε, στον Ατλαντικό λόγω της υπεραλίευσης. Όταν διαπιστώθηκε αυτό, οι αλληλευτικοί στόλοι μετακινήθηκαν πιο βαθιά στον Ατλαντικό. Όταν εκεί λοιπόν εντόπισαν νέα είδη, άγνωστα στην κοινή γνώμη, πάλι κατέληξαν στην υπεραλήψη και αυτό μάλιστα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή για πάνω από 10 χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται νόμιζαν ότι τα αποθέματα θα ήταν ανεξάντλητα, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Για πάρα πολλά από τα ψάρια αυτά δεν έχουμε πληροφορίες ε, ούτε καν για τα βιολογικά τους ε, χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι αυτά είναι ειδικέ κατηγορίες ψαριών. Ορισμένα εξ αυτών ε, ζουν εδώ και 150 χρόνια και πολλές φορές ε, φτάνουν στην φάση της ορίμανσης μετά το 300 έτος, δηλαδή πιο κατηστερημένα και από το ανθρώπινο είδος αλλά εξ αυτών έχουν ε, πολύ χαμηλούς ρυθμούς αναπαραγωγής. Έτσι λοιπόν, τα αποθέματα αυτών των ψαριών άρχισαν να εξαντλούνται. Ένας από τους λόγους που εξαντλήθηκαν ορισμένα αποθέματα είναι ότι δεν υπήρχε κανένας κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, το 2002 ελήφθησαν κάποια μέτρα Καθώς όμως φτάνουμε τώρα πλέον στη φάση όπου ε, πρόκειται να αναθεωρηθεί αυτό το καθεστώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πράγματι το ισχύον καθεστώς ήταν ε, αναποτελεσματικό. Και κατά κύριο λόγο διότι δεν έκανε τη διάκριση ε, ποιος ε, στοχεύει στα αυτά τα ψάρια και ποιος ε, τα αλλιεύει ως παρεπίπτοντα αλλιεύματα. Μπαίνανε όλα στον ίδιο τομέα και γι' αυτό δεν, υπήρχε, δεν υπήρχαν οι σωστοί κανονισμοί ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος ήταν οι ακατάλληλοι εξοπλισμοί. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε τι είδους πρόταση κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό καλούμεθα να συζητήσουμε σήμερα. Η κεντρική ιδέα ε, της πρότασης είναι η εξής. Να μετακινηθούμε από μηχανότρατες ε, ε, τις ε, μηχανότρατες βαθέων υδάτων και απλάδια να περάσουμε στα παραγάδια. Σημαντικό λοιπόν είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο βιώσιμη αλληλεία έτσι ώστε οι αλληλείς να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους ε, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αποφύγουμε ή δυνατόν την πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων. Όλες αυτές βέβαια είναι παραδοχές, ε, τις οποίες καλούμεθα σήμερα να συζητήσουμε. Έχουμε ε, κοντά μας διακεκριμένους επιστήμονες, ε, εκπροσώπους του κλάδου και συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους οποίους ε, θα συζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα πώς ακριβώς μπορεί να γίνει αυτή η ε, μετάβαση. Πιστεύουν πολύ ότι είναι σημαντικό να περάσουμε στα παραγάδια. Ορισμένες χώρες το έχουν ήδη πράξει τα χρησιμοποιούν τα παραγάδια. Άλλοι πάλι λένε ότι το θέμα ε, είναι δευτερεύον. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλήξουμε ως κοινοβούλιο σε θέση. Νομίζω λοιπόν ότι ομιλώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων ε, ισχυριζόμενος ότι όλοι προσβλέπουμε στις εισηγήσεις σας και προσβλέπουμε και σε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Σένη. Ξεκινούμε λοιπόν με το πρώτο πάνελ. Η ανάπτυξη, της, η εξέλιξη της αλληλείας στα βαθιά νερά και ο αντίκτυπός της και δίνω το λόγο στον πρώτο εισηγητή, τον κύριο Τόμ Μπλασντέιλ. Η Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να τηρήσετε 10-11 λεπτά maximum για να υπάρχει και λίγο χρόνο συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Πλάστεϊλ, έχετε το λόγο. Hello, thanks very much picking me up. Okay. Ευχαριστώ. Τον Μπλάσντεϊ λέγομαι. Δουλεύω για την κοινή επιτροπή διαφύλαξης τη φύση του Ηνωμένου Βασιλείου και είμαι πρόεδρο τη ομάδα εργασία του ISIS για την ε, βιολογία και την αξιολόγηση των πόρων βαθιών αλίας βαθαίων υδάτων με το, αρχι... το κρόνιμο WGDEP. Η ομάδα έχει πάνω από 100 ομάδες εμπειρογνωμόνων στο σύστημα του ΆΙΣΕΣ e με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης σε 27 είδη ψαριών στην περιοχή ΆΙΣΕΣ e και να αναφέρουμε τα, ευρήματα στην, Βουλευτική Επιτροπή του ISIS e που παρέχει πληροφορίες στους εμπλεκόμενους όπως τις διοργανώσεις αλλιέων, την διοργανώση διαχείρισης αλλιές και άλλες εθνικές δομές. The slides seem to have got out of order here. Um, okay, there's a lot of missing slides in my presentation. I don't. Λείπουν κάποια slides από την παρουσίασή μου, δεν ξέρω τι έγινε. Okay, well, I have some missing slides, but... Uh, κάποια slides λείπουν. Τέλος πάντων, θα προχωρήσω. Allow me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 θα ανεβάσουμε τη σωστή εκδοχή το συντομότερο δυνατό. Ε, καλά, καλά, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Να σας πω κάτι, κύριε Μπλασδέιλ, μήπως θέλετε να ακούσουμε τον δεύτερο ομιλητή και μετά θέλετε να αλλάξουμε σειρά, λέω κύριε Μπλασδέιλ, σε εσά μιλάω. Adelante. Τέλος πάντων, συνεχίστε, συνεχίστε, ωραία. Right, I'll carry on from here. So what I, what I would like to do in the... Αυτό που θέλω να κάνω είναι να κάνω μια σύντομη εισαγωγή των διαφόρων ε, ειδών αλίας ε, στα βαθιά νερά στην Ένωση και γενικότερα στην περιοχή Άισες με τη δουλειά που έχουμε κάνει για την αξιολόγηση των αποθεμάτων, την κατάσταση αυτή τη στιγμή και κάποια προβλήματα στη διαχείρισή τους. Λοιπόν, τα ίδια αλληλεία στην Ευρωπαϊκή, στα νερά της Ένωσης, από την Ιρλανδική θάλασσα, υπάρχει μεικτή βενθοπελαγική αλληλεία στην περιοχή αυτή, με μια σειρά μεικτών σκαφών ο Γρεναδιέρος, ε, η, ε, η Μουρούνα και σκυλόψερα, αλλά και το σπαθόψερο και το καθευτόψερο του Ατλαντικού με μικρά ποσοστά αλίευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Πιο ανατολικά, στο Κασκαγκεράκι, υπήρξαν, υπήρξε αλία στην περιοχή αυτή στο παρελθόν για Ρεναδιέρο των Βράχων, αλλά αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι πολύ, μικρά τα, ε, πολύ μικρός ο πληθυσμό, Η Ένωση έχει μειώσει το ΤΑΚ ε, και δεν υπάρχει πια αλίευση. Πιο νότια στην Πορτογαλία έχουμε αλίευση για το μαύρο σπαθόψερο και για ε, λιθρίνια στις Αζόρες υπάρχει αλία με διάφορα είδη σε διάφορες φάσεις του έτους, με κυπρίνο και περιτσίδες, ενώ εκτός των υδάτων της Ένωσης στην, ε, στα ανοιχτά του Αταλαντικού υπάρχει μεικτή αλία. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ε, αλλιευμάτων. Η αύξηση της αλλιές ξεκίνησε στο τέλος της δεκαετίας του 80 όταν δεν υπήρχε ρύθμιση της αλλιευτικής δραστηριότητα, τα αλλιεύματα, η αλήθεια στην συνεχίστηκε και στη δεκαετία του 90. Τα στοιχεία που βλέπετε εδώ δείχνουν τις τελικές εκφορτώσεις όλων των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράδειγμα 1 του κανονισμού, όχι στα νερά της Ένωσης, συνολικά στη ζώνη Άισες. Βλέπετε ότι σταδιακά αυξήθηκαν οι αλλιεύσεις στη δεκαετία του 90 με ανώτατο όριο γύρω στο 2004. Τότε ήταν η ακμή τους, τότε που υιοθετήθηκε ο κανονισμός της Ένωσης για τα τάξη, τα ίδια αυτά. Έκτοτε η αλλιεύση μειώθηκε λόγω καλύτερης διαχείρισης. Το επίπεδο των εκφορτώσεων τώρα είναι περίπου λίγο, λίγο λιγότερο από το μισό από το ανώτερο ποσοστό. Σε κάποια αποθέματα, παρότι όπως σας είπα ξεκίνησε γενικά η αλίευση στο, στις αρχές δεκαετίας του 80, υπήρχαν κάποια είδη στα τα οποία είχαμε αλίευση ήδη στο παρελθόν, από τη δεκαετία του 70. Μεταξύ άλλων το σπαθόψαρο στην Πορτογαλία που αλλιεύεται πάνω από 100 χρόνια με παραγάδια. Τώρα, τι συμβουλές έχει παρέσχει η ΆΙΣΕΣ. Ξεκινήσαμε περίπου 10 χρόνια πριν, όταν είχαμε πολύ μικρά, πολύ λίγα στοιχεία για τις εκφορτώσεις. Τα περισσότερα ήταν εξαιρετικά βασικά για κάποια είδη, για μεικτά είδη. Ε, η χρονική περίοδος δεν ήταν ε, σύντομη γιατί δεν είχαμε στοιχεία εποπτείας, ενώ οι βιολογικές πληροφορίες που είχαμε ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Δεν ξέραμε, ας πόσα, την, ηλικία ή την ε, ηλικία αναπαραγωγής των ε, κάποιων ειδών. Και δεν ξέραμε κατά πόσον η, η κατάσταση αλίευσης τότε επέτρεπε την αναπαραγωγή. Έκτοτε, για τα περισσότερα είδη που παραμένουν ε, στην κατηγορία των ε, χαμηλής ε, παροχής στοιχείων δεν μπορούμε να δώσουμε προβλέψεις, αλλά για τα περισσότερα έχουμε κάποια στοιχεία με, με σειρά ετών για ορισμένα από αυτά με αποτέλεσμα να υπάρχει μία αναλυτική αξιολόγηση για τρία είδη. Για τα άλλα δώσαμε καλύτερες πληροφορίες για την, ε, τον έλεγχο της ε, ε, αλίευσης. Πέρσι δώσαμε συμβουλές για τα 27 είδη που καλύπτονται. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα τώρα των ειδών που αξιολογούμε. Πρώτον, για την ε, μουρούνα, την μπλε μουρούνα στις περιοχές που βλέπετε. Αν δείτε το γράφημα επάνω αριστερά, το ίδιο που σας έδειξα και προηγουμένως, δείχνει στις δεκαετία του 70 μεγάλο όγκο αλίευσης, μια δεύτερη ανάκαμψη των, ε, στη δεκαετία του 90 με έναν ανώτατο όριο το 2001, ενώ μετά σταδιακά η αλίευση μειώνεται σταδιακά αφού υιοθετήθηκαν τα μέτρα διαχείρισης. Επάνω δεξιά, το γράφημα πάνω δεξιά, είναι η παραγωγή που έχει γίνει, η, ευθύ, η σταθερή γραμμή είναι ο αριθμός των, ε, ο πληθυσμός. Βλέπετε ότι ο αριθμός στη δεκαετία του, 50, του 90 έφτασε το 1 πέμπτο στην πραγματικότητα του συνόλου και σταδιακά με το 2006 να αυξάνεται. Το, κάτω, κάτω, το γράφημα κάτω δεξιά δείχνει το αντίστοιχη εικόνα μείωση, σημαντική μείωση με μια σταδιακή ανάπτυξη. Κάτω αριστερά είναι η θνησιμότητα του πληθυσμού. Το 2000, στη δεκαετία του 2000 η εθνισμότητα ήταν υψηλότερη και έκτοτε μετά από μέτρα διαχείρισης μειώθηκε σημαντικά και είναι τώρα χαμηλότερα από το επίπεδο αναπαραγωγής. Τώρα η μουρούνα αναπαράγεται γρήγορα, στα 15 χρόνια περίπου, οπότε συνηθίζει, μάλλον μοιάζει με άλλα είδη που βλέπουμε στα, στην υφαλοκρηπίδα. Ένα άλλο και υπάρχει μια δυνατότητα ανάκαμψης του είδους αυτού αρκετά καλή. Το δεύτερο ε, παράδειγμα είναι ο γραναδιέρος των βράχων. 6, 7, 5β και 12β περιοχές. Βλέπετε ότι οι εκφορτώσεις στο είδο αυτό ξεκίνησαν στη δεκαετία του 80, έφτασαν το το όριο στην αρχή της δεκαετίας του 2000 και μετά μειώθηκαν σημαντικά μετά από το καθεστώς διαχείρισης της Ένωσης. Επάνω δεξιά το CPUE δίνει το επίπεδο, το συντελεστή ε, Κάτω αριστερά είναι το επίπεδο θνησιμότητας στην πραγματικότητα, το επίπεδο ε, άντλησης το λέμε, γύρω στο 2007 ήταν η χειρότερη χρονιά, έκτοτε μειώθηκε στο επίπεδο που παρέχει τη μέγιστη εγγυημένη απόδοση ή λίγο χαμηλότερα από αυτό. Υπήρξε μια μακρά μείωση στη δεκαετία του 70 και του 80, τώρα έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα 30% ε, της αρχικής της ε, καθαρής βιομάζας του. Τα τελευταία χρόνια κάπως ε, μεγαλώνει, κάπως αυξάνεται. Η ζωή του είναι μεγαλύτερη, είναι 30 χρόνια, οπότε ο, το, ο, βαθμός ανάκαψης είναι αργότερος. Το τρίτο παράδειγμα, με λιγότερα στοιχεία όπως θα δείτε, το μαύρο σπαθόψαρο. Και εδώ έχουμε αύξηση στη δεκαετία του 80, απνότατο όριο γύρω στο 2000, μείωση ως αποτέλεσμα καλύτερης διαχείρισης. Τα στοιχεία που έχουμε για την αξιολόγηση ε, του αποθέματος είναι το, η αλήψη αναμονάδα προσπάθειας. Μετά βλέπετε ότι εκεί υπάρχει μια σταθερότητα, μια αύξηση στο ξεκίνημα, σταθερότητα και τα τελευταία χρόνια μια μικρή αύξηση. Η γενική εικόνα για τα βενθοπελαγικά Ήδη είναι ότι πολλά από τα ίδια αυτά φαίνεται ότι μετά από τα μέτρα διαχείρισης σταμάτησε η φθήνουσα πορεία. Σε κάποιες περιπτώσεις σταθεροποιήθηκε, άλλοτε όχι. Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να δώσουμε ποσοτικούς στόχους, αλλά είναι δυνατό γιατί η θνησιμότητα είναι αρκετά κοντά στην μέγιστη εγγυημένη απόδοση. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι όταν έχεις μεικτή αλλιεύση και συντελεστή εκμετάλλευση κοντά στο μέγιστο, στη μέγιστη εγγυημένη απόδοση, θα φτάσει σε σημεία όπου είναι οριακά για κάποια από τα λιγότερα παραγωγικά είδη του συστήματος. Η κατάσταση αυτή δεν αφορά μόνο τα, τα είδη της, ε, του βυθού αλλά και, τα επιφανειακά. Για παράδειγμα το κεντρόνι, άλλα είδη καρχαριών που βρίσκονται σε, σε πολύ χαμηλό επίπεδο αναπαραγωγής γιατί ε, τα, μαζε, τα πιάνουν σε μεικτή αλίευση μαζί με άλλα είδη. Τώρα, στην αλία που μας αφορά, στο βαθιά νερά, μεταξύ των ε, πιο ευάλωτων ε, ειδών είναι τα ε, σκυλόψερα. Ποια είναι η λύση τώρα. Πρώτον, να βάλουμε τάκ μηδέν για τα πιο ευάλωτα είδη. Στην Ένωση υπάρχει μηδενικό τάκ για τα σκυλόψερα. Αυτό θα οδηγούσε ωστόσο στην απόρριψη των ειδών αυτών. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις, ε, τα ποσοστά εκμετάλλευση σε επίπεδα που θα είναι τόσο χαμηλά που θα επιτρέπουν να υπάρχει εκμετάλλευση των ευάλωτων ειδών ε, σε βιώσιμο επίπεδο που σημαίνει ότι κάποια από την απόδοση των εμπορικών δραστηριοτήτων θα την αφήνουμε κατά μέρο, θα την εγκαταλείπουμε, ή να υπάρχουν ε, μορφές ε, αλίευσης που θα επιτρέπει να χρησιμοποιούνται τα αλλιευτικά εργαλεία σε συγκεκριμένες περιοχές. Άλλο παράδειγμα ευάλωτων ε, ειδών είναι το καθρεφτόψερο του Ατλαντικού. Και εδώ βλέπουμε ότι στην αρχή της δεκαετίας του 90 η αλίευση πέρασε από το 0 στα 3.500 τόνους και μια ταυτόχρονη μείωση της αλίας όσο αυξανόταν η εκμετάλλευση. Το, το είδος αυτό είναι εξαιρετικά ευάλωτο γιατί είναι είδος με μικρό ρυθμό αναπαραγωγής και μακρά ζωή. Αυτό δείχνει ότι αναείδος χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση της βιώσιμης ε, διαχείρισης. Σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή θα πρέπει να έχουμε εικόνα μιας πολύ μακροχρόνιας ε, εκμετάλλευσης, όχι κάποιων ετών μόνο. Γενικά συμπεράσματα. Πρώτον, η θνησιμότητα των βασικών ειδών έχει μειωθεί σε επίπεδα που είναι είτε κοντά είτε λίγο χαμηλότερα από τα επίπεδα που επιτρέπουν μέγιστη εγγυημένη απόδοση. Τα περισσότερα εμπορικά είδη είναι σταθερά, στον, ο, ο πληθυσμός είναι σταθερός ή αυξάνεται. Κάποια από αυτά τα είδη έχουν σχετικά ταχεία ε, αναπαραγωγή και άρα μπορεί να κτίσουν ε, γρήγορα τον παλιό ρυθμό. Κάποια είδη παραμένουν σε υπερβολική εκμετάλλευση και χρη, ενδεχομένως να χρειαστούν περαιτέρω μέτρα, φερρυπίν, τα διάφορα είδη καρχαριών που, ε, και σκυλοψάνων που αλλιεύονται παρεπιπτόντως. Άλλα, σε άλλα είδη, όπως Το καθεπτόψαρο μπορούμε να συνεχίσουμε την εμπορική δραστηριότητα χωρίς μείζωνα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής. Ο λόγος στον κύριο Φίλιπ Πούιδερ. Δεν λέω ποιος είναι ο καθένας και τι θέση έχει, διότι το, έχετε τους τίτλους του στην ημερήσια διάταξη, έτσι για να γλιτώσουμε χρόνο, ε, δεν διαβάζω την ε, θέση, του αξίωμα ε, κάθε από τους ομιλητές. Παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τους ε, χρόνους που έχουμε δώσει για να γίνει και συζήτηση μετά. Συζήτηση που είναι σημαντικό τμήμα αυτών των ακροάσεων πάντοτε. Παρακαλώ πολύ, κύριε Ούιβερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Σα ε, σας παρουσιάζω αποτελέσματα δύο μεγάλων project, ευρωπαϊκών project. Ε, εργαστήρια, επιστημονικά εργαστήρια εξέτασαν οικοσυστήματα ε, βαθιών υδάτων. Στο δεύτερο project, μάλιστα, αξιολογήσαμε και τις επιπτώσεις ανθρώπινης δραστηριότητες σε βάθη κάτω των 200 μέτρων πάνω στο βυθό. Καταρχήν προσπαθήσαμε να δούμε Ποιε είναι οι δραστηριότητε που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ε, βυθό. Και πιο συγκεκριμένα το έτος 2005 ε, σε περιοχές ΟΣΠΑΡ ε, ε, ε, κάτω από τα 200 μέτρα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που βλέπετε είναι δραστηριότητες που επηρεάζουν τον, το βυθό Έχουμε πετρελοπηγές, έχουμε αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου, έχουμε τις στράτες ε, βυθού, ε, έχουμε ε, εναπόθεση ραδιενεργών καταλήπων, χημικών όπλων και γενικότερα οπλισμού, καθώς επίσης και καλώδια τηλεπικοινωνία στο βυθό. Προσπαθήσαμε να δούμε τι επιφάνεια επηρεάζει κάθε μία αυτές τις δραστηριότητες. Έχουμε λοιπόν αυτή τη γραφική παράσταση. Αριστερά θα δείτε ότι ορισμένε αυτέ τι δραστηριότητε επηρεάζουν πολύ μικρέ επιφάνειε. Δεξιά όμω βλέπετε ότι έχουμε δύο δραστηριότητε οι οποίε ε, έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση. Μία από αυτέ ε, βγαίνει και από την κλίμακα. Έχουν και οι δύο σχέση με τι στράτε βυθού ε, και τα ίχνη του. Έχουμε δύο μπάρε εδώ. Μία για την ελάχιστη και μία τη μέγιστη επιφάνεια, επειδή ακριβώ δεν έχουμε πλήρη στοιχεία. Ξέρουμε όμως ότι η αριστερή μπάρα είναι το ελάχιστο και η δεξιά είναι το μέγιστο σε ό,τι αφορά την επιφάνεια την οποία, ε, στην οποία έχουν επιπτώσεις ε, αυτές οι δραστηριότητες, αυτή η δραστηριότητα συγκεκριμένα. Όπως θα δείτε η επιφάνεια αυτή είναι μεγαλύτερη από το σύνολο όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Ακόμα και αν πάρουμε το ελάχιστο ε, της ε, επιφάνειας την οποία επηρεάζει η αλήψη με τράτες βυθού. Έχουμε ένα Παράδειγμα, ε, ε, με στοιχεία από το 77 μέχρι το 89 όταν δεν η χώρα καμία αλληλευτική δραστηριότητα ε, καταγράψαμε λοιπόν όλα τα, τα είδη τα οποία είχαν εμφανιστεί τότε, είχαν εντοπιστεί τότε. Μετά μου ξεκίνησε η αλίευση και συλλέξαμε τα ίδια στοιχεία μετά από κάποια χρόνια αλίευσης. Και μπορούμε να συγκρίνουμε. Τα, τα κόκκινα, κόκκινες στιγμές είναι τα ε, παλιότερα ε, και οι μαύρες είναι ε, τα νεότερα στοιχεία. Εδώ βλέπετε ένα περίπλοκο γράφημα με τις συνέπειες της αλίευσης. Η μαύρη γραμμή αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες πριν ξεκινήσει η αλίευση. 25.000 ψάρια ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο ήταν η πυκνότητα. Η κόκκινη γραμμή δείχνει τις επιπτώσεις της αλίευσης με μείωση του πληθυσμού σε λίγο παραπάνω από 7.000 ψάρια ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Ε, αλίευση από τα 500 έως τα 1.500 μέτρα περίπου. Αυτή είναι η κατακόρυφη γραμμή την οποία βλέπετε, είναι στα 1500 μέτρα. η επιπτώση, η μείωση δηλαδή της πυκνότητα των ψαριών ε, δεν σταμάτησε όμως στα 1500 μέτρα παρόλο που η αλήψη σταματούσε στα 1500 μέτρα. Συνεχίστηκε μέχρι τουλάχιστον τα 2.500 ε, μέτρα βάθος. Για να μην σας πω στις 3.000 όπου οι ε, συνεχείς στέμνονται. Συνεπώς ε, οι επιπτώσεις ε, ξεπερνούν τις, ε, το, τα βάθη στα οποία γίνεται η αλίευση. Εδώ βλέπετε το λόγο. Αριστερά βλέπετε το βάθος, η κλίμακα του βάθους, ο κατακόρυφος άξονας. Ε, οι κατακόρυφες γραμμές που βλέπετε είναι όλα τα είδη τα οποία ζουν σε αυτές τις περιοχές και ζουν πολύ κοντά στο βυθό. Πολλά από αυτά ζουν βέβαια σε πολλά βάθη. Ένα από αυτά φτάνει, ε, ζει σε, από λιγότερο από χιλιά μέτρα μέχρι τα 5.000 σχεδόν μέτρα. Συνεπώς ε, όλα αυτά μετακινούνται. Ε, το, η μπλε γραμμή είναι το βάθος στο, στο οποίο γίνεται αλίευση, η μπλε ζώνη. Οτιδήποτε μπαίνει σε αυτή τη ζώνη 500-1500 μέτρα, ε, είναι δυνατόν να αλλιευθεί. Συνεπώ, παρόλο ότι αλλιευόντουσαν μόνο 4-5 εμπορικά είδη, στην πραγματικότητα συναλλιευόντουσαν 78 ε, σχεδόν, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα είδη. 78 συνολικά. Συνολική επιφάνεια ε, η οποία, στην οποία υπάρχουν επιπτώσεις είναι ε, όχι η κίτρινη στην οποία γίνεται η έλλειψη, αλλά η κόκκινη που είναι τρεις φορές ε, περισσότερη. Δηλαδή η κίτρινη και η κόκκινη μαζί είναι 142.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μόνο η κίτρινη που γίνεται η αλήψη είναι 52.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μετά κάναμε μια χαρτογράφηση, Νορβηγία για παράδειγμα, όπου βλέπουμε ε, πολλούς κοραλιογενείς υφάλους. Ο κάθε κόκκινη στιγμή κάθε κόκκινο σημαδάκι είναι ένα κορολογενή ύφαλο. Ε, είναι δεκάδες μέτρα μήκο έχουν έχει καθένας από αυτού. Ε, δεν μιλούμε μόνο για κοράλια όμω, ε, διότι υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα εκεί στα κορολογενή ύφαλου. Ε, είναι πολύ περίπλοκη λοιπόν η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολη η χαρτογράφηση εκτός και αν έχεις πολύ ακριβό εξοπλισμό και υψηλή ευκρίνεια. Ε, Παρ' όλα αυτά, ο κανόνα ε, τη μετακίνηση, το οποίο σημαίνει ότι η Αλία θα πρέπει να μετακινείται μακριά ε, από κορολογενεί υφάλου κλπ. Ε, αν αλλιεύει ε, κάποιε ποσότητε σουγκαριών ή κοραλιών μεγαλύτερε από ένα όριο. Ε, Αυτό είναι ο κανόνα, αλλά πόσο μακριά θα πρέπει να μετακινηθεί. Δύο ναυτικά μίλια από εκεί που εντοπίζεται πίστηκε το οικοσύστημα. Οπότε αν κάπου σε ένα ίχνος εντοπίσει κοράλια, η μετακίνηση κατά δύο ναυτικά μίλια σε ρίχνει πάνω σε ένα άλλο ίχνος, όπως βλέπετε διακεκομένες μέσα εδώ, το οποίο σημαίνει ότι ενδεχομένως η μετακίνηση να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα, διότι μπορεί να, με τη μετακίνηση να αρχίσεις να επηρεάζει πολύ περισσότερες διακεκομένες γραμμές, όπως βλέπετε σε αυτό το διάγραμμα. Οπότε, ε, επίσης, τίθεται θέμα του πώς συλλέγουμε επιστημονικά στοιχεία και πόσο περίπλοκο είναι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ενός, μιας ε, αποστολής που κόστησε 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Γενογραφικό Ινστιτούτο του Βασιλείου το 2011 ε, χαρτογράφησαν ε, μια μικρή επιφάνεια βυθού και μετά με κάμερες και ε, εξοπλισμό χαρτογράφησης μέτρησαν τις επιπτώσεις της αλίευσης στην περιοχή όχι μόνο που γινόταν αλίευση αλλά σε μια πιο ευρεία περιοχή. Αν δούμε λοιπόν ε, εδώ ε, βλέπετε έχουμε ε, μια μικρή περιοχή αλίευσης η οποία χαρτογραφήθηκε βλέπετε είναι σαν ένα ορθογώνιο και μια ευρύτερη περιοχή. Τα τρία μαύρα τετραγωνάκια αντιπροσωπεύουν στοιχεία υψηλής ευκρίνειας με, ιδιές, με ειδικές κάμερες βυθού. Τα εσωτερικά κουτιά μέσα στο ΜΟΒ στη περιοχή, είναι περιοχές προστασίας, προστατεύονται από την αλλιεύση και ε, έχει γίνει πρόταση να, ε, ε, να επεκταθούν στο, να, ώστε να καλύψουν όλο το πράσινο κομμάτι. Ε, εδώ βλέπετε δύο φωτογραφίες. Η ε, πρώτη, ε, πρώτη είναι αυτή με το οικοσύστημα το οποίο είναι ανέγγιχτο στο, μέσα στην περιοχή που προστατεύεται με κοράλια, πολλά ψάρια και άλλους οργανισμούς. Αν το δούμε από κοντά θα, θα φανεί αυτό. Και εδώ είναι ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά τα ψάρια αυθονούν, αναπαράγονται κλπ. Είναι μια υγιής κοινότητα. Ε, είναι μια περιοχή που πρέπει να προστατευτεί. Είναι ένα οικοσύστημα χρήσιμο και υγιές. Στην άλλη περιοχή, εκεί που προτείνεται να γίνει επέκταση, βλέπουμε αυτό. Είναι ένας νεκρός βυθός, κομμάτια κοραλιού, ο, ίχνη από τράτες που πέρασαν αυτή η περιοχή θα πρέπει να είναι ίδια με την προηγούμενη φωτογραφία. Όμω έχει καταστραφεί από τράτα. Ούτε έχουν μείνει βέβαια ψάρια. Οπότε όλη η, η κοινότητα έχει εξαφανιστεί. Αυτό ανησυχεί του επιστήμονε γιατί θα χρειαστούν χιλιάδε χρόνια για να αναγεννηθεί. Τα βασικά συμπεράσματα. Ε, οι μηχανότρατες ε, βυθού έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Βυθού πολύ περισσότερο από όλες οι άλλες δραστηριότητε μαζί. Δεύτερον, η αλίευση ε, μεγάλα βάθη έχει ένα δυσανάλογο, μια δυσανάλογη, έχει δυσανάλογη σε είδη τα οποία δεν είναι εμπορικά και επηρεάζει και περιοχές εκτός της ε, περιοχής αλίευσης. Ε, υπάρχουν ε, μέτρα για να αποφευθεί αυτή η καταστροφή, αλλά δεν είναι αρκετά και ενδεχομένως καταστρέφουν περισσότερα Ε, Επίσης τα, τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε δεν είναι αρκετά. Η, περιοχή, η κατάσταση είναι περίπλοκη και θα πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ. Τελείωσε η, το πρώτο πάνελ. Ας κάνουμε ένα πρώτο γύρο που παρακαλώ να μην είναι σκέψεις και παρατηρήσεις αλλά συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους ηγητές. Ο κύριος Στίβενσον πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους δύο ομιλητές, τον κύριο Μπλάσντερ και τον κύριο Γουίβερ για τις παρουσιάσεις τους. Υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ των δύο παρουσιάσεων, έχω την εντύπωση. Αφενός, η ISIS μας λέει ότι σε πολλά είδη τα μέτρα διαχείρισης οδήγησαν σε ανάσχεση της ιστορικής ε, φθήνους και ότι σε κάποια είδη υπήρξε αύξηση των αποθεμάτων. Κατόπιν όμως έχει το κύριο Βίβερ και μας λέει ότι πρέπει να, σταμα... να, να κλείσουμε συγκεκριμένες περιοχές από οποιαδήποτε μορφή αλίευσης που θα έχει προφανώς κοινωνικές επιπτώσεις για τους ε, ψαράδες και τις οικογένειές τους. Εγώ είχα ανέβει κάποτε σε μια τράτα που είχε προσαρμοστεί για αλία σε βαθιά νερά, στη Σκοτία, που είχαν κάνει σημαντικές επενδύσεις για να αλλάξουν ε, το σκάφος προς το σκοπό αυτό. Φαντάζομαι ότι παρόμοια δουλειά θα έχουν κάνει και πολλά σκάφη άλλα στην Ευρώπη. Εκτιμώ λοιπόν την ευαισθησία για τα ίδια αυτά που έχουν μακρά περίοδο ορίμανσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους ψαράδες. Με ενδιαφέρουν και οι άλλες, και άλλες παρουσίες, αλλά το να ξεκινάμε στην ακρόαση αυτή με προτάσεις για πλήρη απαγόρευση δεν βοηθάει. Θα ήθελα να συζητήσουμε μετά την αντίφαση που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών ε, ε, παρουσιάσεων. Ο κύριος Ρωμέβα. Πολλές ερωτήσεις, αν κατάλαβα καλά. Το μήνυμα που περνά από τον κύριο Μπλάσντελ βασικά είναι η προφανής κατάσταση των επιπτώσεων της μικτής αλίευσης. Η ερώτηση είναι απλή. Και όταν έχετε μεικτή αλία, ανεβάζεις τα τάκ για κάποια είδη. Οι συνέπειες όμως για τα πιο ευάλωτα είναι πολύ πιο δυσδιάκριτοι. Δεν μπορείς να τους προστατεύσεις. Και μηδέν τάκ να βάλεις για το σκυλόψαρο, αν το πιάσεις ως παρεμπίπτον, έχεις ένα πρόβλημα ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δεύτερον, αφελής ίσως η ερώτηση. Είπατε συχνά, μιλήστε συχνά, για, για την έλλειψη στοιχείων ή για ανεπαρκή στοιχεία. Γιατί πού έγκυται τα προβλήματα της κτήσης πληρέστερων στοιχείων. Και προς τον κύριο Βίβερ. δύο ερωτήσεις και εκεί. Ο κλάδος επανειλημμένα ανέφερε ένα βασικό μειονέκτημα. Την αλίευση με τράτες βυθού. Η ερώτηση που θέτω είναι η εξής. Εγώ είδα τον αντίκτυπο και τη ζημιά που κάνει ένα συγκεκριμένο είδος αλίευσης. Εσείς τι άποψη έχετε. Γιατί δίνουμε τόση έμφαση μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη μορφή αλίας. Πέραν του αντικτύπου που έχει η αλία, υπάρχουν συνέπειες Λοιπόν, ποιος είναι ο αντίκτυπος για την παρούσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Τωμά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ στους εμπειρογνώμονες. Ένα μια ερώτηση στον κύριο Βίβερ. Στο, στην Nature το 2012 ε, δημοσίευσατε τρεις χαρακτηριστικές ζώνες ε, με στοιχεία ε, όπως αυτά που μας δείξατε, με επιπτώσεις ε, λόγω μεγάλης αλίευσης ε, με μια περιοχή με μέτρια ε, αλίευση και μια περιοχή που θα πρέπει να γίνουν περισσότερες έρευνες. Αυτές οι διαπιστώσεις δεν μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να έχουμε διαφορετικές ζώνες. Υπάρχουν ζώνες που έχουν υποστεί πολύ αλίευση και έχουν χειροτερεύσει πολύ συνεπώς δεν θα ανασυσταθούν, ε, οπότε ε, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την αλλιεύση εκεί, αλλά και άλλες ζώνες που είναι σε καλή κατάσταση και εκεί θα πρέπει να τις προστατεύσουμε. Και δεύτερον, τον κύριο Μπλαστέιλ. Για τα ευαίσθητα ευάλωτα είδη αναφερθήκατε. Οπότε σε συνάρτηση με τη χρήση αυτών. Ε, σχετικά με τους καρχαρίες υπάρχει περίπτωση τα σκυλόψερα δηλαδή να επιβιώσουν έτσι όπως είναι η κατάσταση. Νομίζω ήταν και οι δύο πολύ καλές οι παρουσιάσεις. Θα συμφωνούσα με τον κύριο Στίβενσον. Ε, η μία φαινόταν να είναι αισιόδοξη ενώ η άλλη απεσιόδοξη. Θα ήθελα να μου εξηγήσουν δύο μιλητές αυτή τη διαφορά το καθρεπτό ψαρό. Είναι πολύ κλασική περίπτωση. Πόσα εκατοντάδε χρόνια χρειάστηκε να ε, αυξηθεί ο πληθυσμό τόσο πολύ και μετά σε ένα χρόνο αλίευση εξαφανίστηκαν. Δεν είναι δυνατόν να ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι το κλασικό παράδειγμα του τι κάνουν οι άνθρωποι στον ωκεανό. Έχω όμω μία ερώτηση για τον κύριο Βίβερ. Μα δώσατε ένα κατάλογο ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και επιπτώσεων του. Μία ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν αναφέρατε ήταν οι ανεμογεννήτριες ε, ανοιχτής θαλάσσης. Οι ψαράδες λένε ότι γύρω από τέτοιου ανεμογεννήτριε, ανεμογεννήτρες 500-500 μέτρα απόσταση δεν βρίσκεται ούτε ένα ψάρι. Ισχύει αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σκαντέκ. Euh, Ευχαριστώ στον κύριο Πλαστέλ και στον κύριο Βίβερ για την ποιότητα των παρουσιασεών Όπως είπε ο κ. Στίβενσον, ε, εντόπισα ορισμένε αντιφάσεις, νομίζω και οι υπόλοιποι, ανάμεσα στις ε, δύο παρουσιάσεις. Για ένα τμήμα των όσων είπαν τουλάχιστον. Με εντυπωσιάζει επίσης ότι ο κ. Μπίβερ η, η κύριο Βίβερ, η το πρώτο τη παρουσιασή σα σταματούσε το 2005, αν δεν κάνω λάθο. Ε, το τέλος, στο τέλο τη σας, σα, λίγο πριν το τέλος, μας δείξατε τις ακτές που δεν νομίζω ότι έχουν άμεση σχέση με τον τομέα τον οποίο ε, ε μελετούμε σήμερα. Μετά ο κύριος Μπλάσδελ μας είπε ότι τα αποθέματα είναι σε καλή κατάσταση και μάλλον έχουν τάση ανασύστασης. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, αυτό άκουσα. Όπως είπε ο κύριος Στίβενσον, αντί να μιλήσουμε για πάυση δραστηριοτήτων, θα πρέπει να μιλήσουμε για καλή διαχείριση. Και μία ερώτηση και προς τους δύο. Ε, τι πιστεύει ο ένας για τον άλλον. Ε, τι πιστεύετε μάλλον ο ένας και ο άλλος ε, για την αρχή του παγώματος που θα επέτρεπε μια καλή διαχείριση αντί για πλήρη απαγόρευση. Ευχαριστώ. Sí, quería también agradecer a los dos intervinientes y quería hacer una... Κυρία Φράγα, έχω μια σειρά ερωτήσεων. Κύριε Ούιβερ. Κύριε Ούιβερ, λοιπόν. Ε, διακρίνατε ανάμεσα στις επιπτώσεις μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων. Ε, προφανώς ε, δεν είναι όλα τα οικοσυστήματα ίδια. Συνεπώς και οι επιπτώσεις δεν μπορεί να είναι οι ίδιες άλλο μια, ένας αμμώδης ε, ε πυθμένας και άλλο ένας πυθμένας με κορεράλια. Έτσι, κάνατε διάκριση ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους πυθμένα βυθού. Δεύτερον, πώς μετρήσατε τις επιπτώσεις κάθε μιας από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα ήθελα να μου πείτε πώς μετρήθηκε ο, αντίτυπος, ο αντίκτυπος. Λέτε ότι οι επιπτώσεις του, της ε, αλήψης μετράτες ε, βυθού είναι πιο μεγάλες. Αλλά πώς μετρήθηκαν. Τρίτον, υπάρχει μια αντίφαση Η, η έκθεση Deep Frisman αναφέρει ότι είναι δυνατόν να πάρουμε και άλλα στοιχεία με κόστος πολύ χαμηλό. Μιλήσατε για το κόστος των στοιχείων, έτσι. Ε, η Deep Frisman ε, λέει ότι υπάρχουν τρόποι ε, να, να πάρουμε στοιχεία με χαμηλότερο κόστος. Μετά, μία ερώτηση και προς τους δύο. Ε, μιλούμε για μια πρόταση της Κομισιόν που θέλει να παγορέσει πλήρως ε, τις, ε, τις στράτες βυθού. Είναι προφανές ότι δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ζουν το ίδιο όλα τα είδη, αλλά αναπαράγονται πιο γρήγορα, μεγαλώνουν πιο γρήγορα κλπ. Ε, τούτου λεχθέντος και ε, λαμβάνοντας υπόψη ως επικαιός Σουίβερ θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, εστιαστούμε σε ευάλωτα οικοσυστήματα με κανόνες ακόμη πιο αυστηρούς από αυτούς που έχουμε, ε, περιοχές απαγόρευσης, αλίευσης ε, ή περιοχές ε, που θα εφαρμόζουν τον κανόνα μουβών της μετακίνησης, δηλαδή με πιο αυστηρό τρόπο ή με ειδικά μέτρα για συγκεκριμένα είδη, δεν θα ήταν αρκετό δεδομένων των αποτελεσμάτων που έχουν δώσει τα μέτρα διαχείρισης από το 2004. Γιατί ε, με την πρόταση της ε, Κομισιόν είναι σαν να σκοτώνουμε μύγες με κανόνια. Γιατί ε, σε περιοχή ναύκων, νεάφ και κοινοτικών υδάτων ε, οι επιπτώσεις δεν έχουν μετρηθεί από την Κομισιόν αλλά οι οικονομικές και οι κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλες μιλάμε για βιώσιμότητα, κοινωνική, οικονομική κλπ. Θα πρέπει να λαμβάνουμε και τα δύο πράγματα υπόψη. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας άποψη. Ε, μήπως εστιαζόμασταν στα ευάλωτα οικοσυστήματα που συστήνουν και οι θα τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΦΑΟ με τις ε, κατευθύνσεις γραμμές τους. Δεν θα ήταν αρκετό. Ευχαριστώ κύριε Φράγκα. Ευχαριστώ. Η προσέγγιση των δύο εισηγητών που ευχαριστώ για τη διαφάνεια και για τη σαφήνεια της παρουσίασής του ήταν τόσο αντιφατική όπως ε, πιστεύουν οι περισσότεροι από εσά. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν δύο αντιμαχόμενες ε, αλήθειες και ότι το ένα είναι αλήθεια και το άλλο ψέμα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι απεσιόδοξοι οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Ο κύριος Μπλάσντέιλ ε, μελετά εμπορικά είδη ξεχωριστά. Και αδιαμφισβήτητα έχει στοιχεία για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό ή εκείνο το είδος σταθεροποιήθηκε τουλάχιστον ως προς την αναπαραγωγή, την ανανέωση. Ο κ. Βίβερ, αντίθετα, εξετάζει τις επιπτώσεις της αλίας στο σύνολο του 20, στο συνολικό οικοσύστημα και σε άλλα είδη. Εγώ είδα ένα νούμερο που με εντυπωσίασε για 4-5 εμπορικά είδη υπάρχουν άλλα 75 τα οποία απορρίπτονται. Αυτές είναι δύο μέθοδοι Ποια από τις δύο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στις μελέτες. Προφανώς δεν μπορούμε να απορρίψουμε τη μία ή την άλλη. Η ερώτηση που θέτω στον κύριο Ντέιλ είναι το Συμβούλιο Υπουργών πρόσφατα, το Δεκέμβριο νομίζω, στηρίχθηκε μόνο στην, στην, ανάλυση, στην ανάγνωση μάλλον της ε, ανανέωσης των αποθεμάτων βαθιών υδάτων για να αυξήσει σημαντικά τις ποσοστώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους ε, όσοι ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία το να έρθουν οι εμπειρογνώμονες και να μας ε, ενημερώσουν για την κατάσταση σχετικά με τα είδη βαθέων υδάτων. Βεβαίως ε, θα ήθελα να γνωρίζω ε, κατά πόσον υπάρχουν ε, ψάρια ε, των οποίων εξαντλούν τα αποθέματα και άλλα που εμπλουτίζουν τα αποθέματά τους σε περίοδο κάτω των 15 ετών. Η Μουρούνα κάτω των 15, ο Γραναδιέρος άνω των 30. Ε, θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζουμε το χρονικό διάστημα και μετά ε, συγκεκριμένα να στοχεύσουμε σε αυτά τα είδη βαθέων υδάτων. Gracias, señora, Κύριε Αρσένης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρέπει να πω ότι με σοκάρισαν, με εντυπωσίασαν και οι δύο ομιλίες. Κυρίως η ομιλία του κυρίου Μπλάστελ. Στο γράφημα μπορέσαμε να δούμε πόσο γρήγορα εξαντλήθηκε το απόθεμα πρέπει να πω ότι πραγματικά ε, σοκαρίστηκα. Νομίζω υπάρχουν κάποιες ε, παρεξηγήσεις. Θα ήθελα να έχω μία σαφή εικόνα. Σχετικά με τα τάκ που προτείνονται. Ποια είναι τα αποθέματα που αυξήθηκαν, πόσα μειώθηκαν, ποια παρέμειναν ε, μηδενικά και ποια αποθέματα παρέμειναν σταθερά. Αυτά θα ήθελα να γνωρίζω. Ας δώσουμε το λόγο στους δύο προσκαλεσμένους μας που έχουν πολλές ερωτήσεις να απαντήσουν. Παρακαλώ πολύ όμως σύντομα, γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές και πολλή συζήτηση μπροστά μας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει, όποιος από τους δύο επιθυμεί. Señor Weaver, okay, okay. Let, let me just try to clarify this issue about... Um... Weaver. Να σας διευκρινίσω λίγο τις ε, διαφορές μας. Έχουμε τρεις ε, διαφορετικές κουτύπου επιπτώσεις. Πρώτον, στα είδη τα οποία αλλιεύονται, αυτά για τα οποία μίλησε ο κ. Μπλαστέιλ, έχουμε επιπτώσεις σε άλλα είδη, τα οποία αλλιεύονται, που δεν είναι όμως αυτά που ήταν ο στόχος των αλλιών, και μετά έχουμε επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα οικοσυστήματα κλπ. Και γι' αυτό εγώ μίλησα για αυτό το τρίτο, είδο επιπτώσεων, αυτό είδος επιπτώσεων κυρίως. Και για το δεύτερο, αλλά λιγότερο. Δεν είμαι κατά της αλίευσης. Απλά θέλω να μπορώ να δω το μέλλον των παιδιών μου και των εγγονιών μου και ως αλλιών και ως ανθρώπων που θα τρώνε ψάρι. Συνεπώς είμαι υπέρ της αλίευσης με σεβασμό του περιβάλλοντος. Αν μπορούσαμε να αλλάξουμε τις πρακτικές αλίευσης έτσι ώστε να πετύχουμε την βιωσιμότητα, πολύ ευχαριστώ. Ε, Είπα ότι μιλώ για περιοχές κάτω των 200 μέτρων, μεγαλύτερο βάθος από 200 μέτρα. Ε, δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες εκεί ε, δεν θα μπορούσαμε, δεν είχαμε αρκετό προπολογισμό ε, να, για να δούμε και περιοχές με βάθος επιθυμένα κάτω των 200 μέτρων. Ε, για το θέμα των νορβηγικών ακτών. ήταν βαθιά ύδατα στα ανοιχτά της Νορβηγίας. Ήταν παράδειγμα περιοχών που υπάρχουν κοράλια. αλλού έχουμε πολύ μεγάλες περιοχές με κοράλια, και αλλού ε, μικρές συστάδες κοραλιών, ε, κοντά η μία στην άλλη όμως, οπότε θα μπορούσαν ε, να επηρεάζουν πολλές ταυτόχρονα. Τώρα, οι επιπτώσεις κάθε μιας δραστηριότητα και πώς τις μετρήσαμε. Αυτό που κάναμε ήταν ότι προσπαθήσαμε να μετρήσουμε την επιφάνεια βυθού που επηρεάστηκε από κάθε μία από τις δραστηριότητες. Ένας ε, ε, αγωγός φυσικού αερίου πετρελαίου, για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο, ε, τι επιφάνεια βυθού επηρεάζει. Η αλία βυθού επηρεάζει μέσω των ιχνών της μεγάλες επιφάνειες που πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται και εν πάση περιπτώσει υπολογίσαμε πόσο ήταν το 2005. Συνεπώ, το κριτήριο, το μοναδικό μας κριτήριο ήταν η επιφάνεια του πυθμένα που ε, επηρεάζεται. Ε, για τα αποθέματα προφανώς ε, ραδιονεργών καταλήπων κοιτάξαμε και έτη προηγούμενα. Αλλά για τις στράτες μόνο το 2005. Αυτά. Μπορώ να δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο, τον κύριο Βλαστέρη. Ευχαριστώ. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίφαση ή αντίθεση μεταξύ αυτών που είπε ο κ. Γουίβερ και εγώ στις παρουσιάσεις μας. Εμένα, μάλιστα, με εντυπωσία το πόσο κοντά ήταν οι δύο παρουσιάσεις. Αν δείτε τα γραφήματα που σας, έδωσα, που σας έδειξα για την κατάσταση των αποθεμάτων κατά την περίοδο που υπήρχε εξαιρετικά μεγάλη μείωση της αλίευσης, θα διαπιστώσετε ότι σε μερικέ περιπτώσει, οι πληθυσμοί έφταναν το 30% τη αρχικής περίοδου και η πληθώρα αλίας, η διαφορά μάλλον μεταξύ της αλίευσης και της μη αλίευσης μειώθηκε από 25 σε 7 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Υπάρχει μια σοβαρή αντιστοίχηση λοιπόν μεταξύ των δύο ευρημάτων αν δείτε, εμείς βλέπουμε μόνο τα εμπορικά είδη. Εκεί η μείωση ήταν 30% σε σχέση με την νοχικό πληθυσμό. Προφανώς, όταν υπάρχει εκμετάλλευση, εμπορική εκμετάλλευση ενός είδους, θα ελπίζαμε, θα περιμένουμε μάλλον να υπάρχει μείωση του πληθυσμού. Σε πολλές περιπτώσεις, η μεγαλύτερη εμπορική απόδοση ενός αποθέματος είναι όταν είναι στο 50% της ε, αρχική, του αρχικού πληθυσμού. Αυτό είναι το επίπεδο που δίνει ε, τη μέγιστη εγγυημένη απόδοση. Τώρα για την αποκατάσταση. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι όταν σταματήσουμε γίνεται ανάκαμψη, αποκατάσταση. Αυτό που λέμε είναι ότι η εκμετάλλευση ή η οριμότητα βρίσκεται σε ένα επίπεδο αυτή τη στιγμή που επιτρέπει ή που θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάκτηση. Ξέρουμε ότι κάποια είδη ζουν περισσότερο, κάποια λιγότερο. Άρα θα υπάρχει μια μεταβολή, μια, μια μεταβλητότητα στα, στην ταχύτητα της ανάκτησης. Μέχρι τώρα δεν έχουμε επαρκή εμπειρία διαχείρισης των αποθεμάτων αυτών για να ξέρουμε πόσο, σε πόσο καιρό θα γίνει η αποκατάσταση, ή θα γίνει στην πρώτη, σε πρώτη φάση. Εμείς μπορούμε να σας πούμε μόνο πόσο χρειάζεται μία ανάκαμψη σε κάποια είδη και με πολύ χαμηλό επίπεδο θνησιμότητας, καρχαρίες για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιμένετε ανάκαμψη χωρίς περαιτέρω μέτρα διαχείρισης για να μειωθεί περαιτέρω η θνησιμότητα. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Κάποιος ρώτησε τι πρέπει να κάνουμε, να σταματήσουμε την αλίευση ή να βελτιώσουμε τους κανόνες. Αν απαγορευόταν η αλίευση με απλά διαβυθού και πηγαίνουμε στο παραγάδι, θα μειωνόταν ο αντίκτυπος στον πυθμένα. Και μπορεί κάποια είδη να αντιμετώπιζαν ακόμα προβλήματα, αλλά ε, η αλίευση θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ο αντίκτυπος στο περιβάλλον θα μειωνόταν σημαντικά αν υπήρχε παραγάδι και όχι απλά διαβυθού κάποιος ε, βουλευτής ρώτησε για περιοχές όπου υπήρχε αύξηση της αλίευσης και την δημιουργία ζωνών και για το αν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε άψες, οικολογικές ε, και βιολογικές ζώνες προστασίας του πυθμένα. Υπάρχουν κάποια τμήματα του πυθμένα που έχουν βιολογική σημασία δεν είναι περιοχέ όπου απαγορεύεται κάθε είδου ανθρώπινη δραστηριότητα αυτή τη στιγμή. Απλά το, τονίζουμε λίγο και λέμε εδώ θα πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση του τι θα γίνει, γιατί αν κάνετε κάτι εδώ θα έχει αντίκτυπο και αλλού. Σε μια τέτοια πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης μπορεί να δούμε ότι σε κάποιες περιοχές θα πρέπει να περιορίζεται πολύ η αλλιεύση και σε άλλες να απαγορεύεται παντελώς. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι βυθός ή όχι αναγκαστικά. Η δημιουργία ζωνών δεν, έχει, λοιπόν, δεν είναι άμεσα σχετιζόμενη με την προστασία των ειδών. Και κάτι ακόμα ξέχασα. ο αριθμός των ειδών που μειώνονται, ε, παραμένουν σταθερά ή αυξάνονται. Δεν έχω μαζί μου τα στοιχεία. Και δεν είναι εύκολη η απάντηση, γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ελληματική ως προς τα δεδομένα. Σε πολλά είδη δεν έχουμε ακριβή αξιολόγηση των αποθεμάτων με χαμηλά, χαμηλής ποιότητας στοιχεία. η σταθερότητα, η αύξηση, η μείωση των ειδών εξαρτάται και από τη χρονική περίοδο της ε, δειγματοληψίας. Σε κάποια περίπτωση, ας πούμε, βλέπουμε μια ανάκαμψη τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Σε μακροπρόθεσμη εικόνα αυτό μπορεί να δείχνει σταθερότητα. Δεν είναι... Δεν υπάρχει απλή απάντηση στην ερώτησή σας. Τώρα, παραγάδια, απλάδια, Συμφωνώ με τον κύριο, με τον, με τον δόκτωρα Βίβερ. Ο αντίκτυπος της αλίευσης με απλά διαβυθού είναι πολύ σημαντικότερος. Το παραγάδι δεν είναι ότι δεν έχει επιπτώσεις. Συχνά τα παραμαγάδια πηγαίνουν το ένα πίσω, ε, ε, το ένα πίσω από το άλλο, ε, τραβάνε και κοράλια σέρνουν, παρασέρνουν και κοράγια. Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένο είδος των παραγαδιών δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ξέρουμε ωστόσο ότι για τους καρχαρίες αυτό είναι αρνητικό και δηλαδή το να αλλάξουμε ε, τη μορφή αλίας από τα, το βυθό στα παραγάδια να έχει αντίκτυπο στα, ε, στους καρχαρίες συγκεκριμένα. Τελειώσαμε αυτό το πρώτο τμήμα της συζήτησης και ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Προχωράμε στη δεύτερη ομάδα. Το Νερέιντα. Η αλίευση Deep Fishman και Νερέιντα, δύο έργα. Ο κύριος Πασκάλ Λοράν, συντονιστής για το Deep Fishman. 10-11 λεπτάκια εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία του Deep Friesman. Ήταν ένα ευρωπαϊκό εργαλείο με 13 εταίρους από 9 χώρες. 3 εκατομμύρια ευρώ υπολογισμό. είχε με κύριο στόχο την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγηση των αποθεμάτων Biological Reference Points, BRP. Ε, Σα τα λέω αγγλικά γιατί στα γαλλικά δεν υπάρχουν και Harvest Control Rules επίσης. Στρατηγικές διαχείρισης και αξιολόγηση, και ορισμό των αναγκών παρακολούθησης και εποπτείας των αποθεμάτων αυτών. Το Deep Fishman ε, στηρίχθηκε σε πολλές μελέτες περιπτώσεων, τα βλέπετε εδώ. Στην, ακρία, στην ακρόαση αυτή ήδη μιλήσαμε για τα σκυλόψερα και εγώ έβαλα κόκκινα σημείο σε κάποιες περιπτώσεις μελέτης όπου οι, οι αναλύσεις έδειξαν, ε, είχαν επίπτωση και σε σκυλόψερα. Κάτι που και δείχνει ότι και εμάς μας ε, ανησυχεί. Θα σας μιλήσω για κάποιους τομείς όπου το Deep Fishman επέτρεψε να υπάρξει πρόοδος. Πρώτον, στον ορισμό του τι είναι περιβάλλον βαθέων υδάτων και είδη, την εκτίμηση των αλληλευτικών προσπαθειών και τις επιπτώσεις στη διαχείριση, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, καθώς και τις υφιστάμενες τάσεις, μεθόδους αξιολόγηση των αποθεμάτων και εν τέλει Δύο-τρία λόγια για τις εξελισσόμενες δραστηριότητες καθώς και τη μελλοντική έρευνα. Πρώτον, το περιβάλλον ε, του βυθού. Εξετάσαμε για το έργο μας ως περιοχές βαθέων υδάτων τους, τους βιότοπους ε, κάτω από 200 μέτρα βάθος. Είναι γενικά αποδεκτός αυτός ο όρος, αλλά οι καθοδηγητήριες γραμμές του, του σε διεθνέ επίπεδο για την αλία σε βαθιά νερά δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένο όριο βάθους. Εμείς λοιπόν λέμε ω περιβάλλον βαθέων υδάτων ότι είναι βαθύτερο από τα 200 μέτρα. Αυτό είναι ε, σε, ε, ευθυγραμμίστηκε με αυτό που είπε ο κύριος Βουίδερ. Τα είδη τώρα της αλίευσης είναι τα είδη που φτιάξαμε έναν κατάλογο όσο πιο αντικειμενικό γίνεται, με ένα ποιοτικό κριτήριο για να διακρίνουμε μεταξύ των επιφανειακών, των αφρόψερων και των, ε, ναι, και των ψαριών ε, βαθαίων υδάτων. Για μας, ήδη είδη βαθαίων υδάτων είναι όσα πάνω από 5% του πληθυσμού τους βρίσκεται σε, σε επίπεδο χαμηλότερο από τα 200 μέτρα βάθος. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τα είδη που περιλαμβάνονται στα παρατήματα 1 και 2 του υφιστάμενου κανονισμού, της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιοι να προσθέσουμε κάποια είδη όπως τον υπόγλωσσο ή τον ασεβαστό. Έχετε εδώ μία εικόνα του, της φαλοκρηπίδας τελείως έτσι σχηματικά. Βλέπετε τα είδη που ε, για μας είναι αυτά που ε, την χάνουν εκμετάλλευση μεταξύ 750 και 1500 ε, μέτρων. Αυτά είναι τα βασικά είδη. Τώρα, το θέμα της αλλιευτικής προσπάθειας. Δουλέψαμε με κάποια στοιχεία παρακολούθηση σκαφών μέσω δορυφόρου. Τα γραφή, το γράφημα επάνω αριστερά είναι στοιχεία για όλα τα σκάφη που ψαρεύουν με δράγες ε, ή ούτε πάνω οποιαδήποτε είδου στράτα στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη βοήθεια των ε, συναδέλφων από το ΣΥΦΑΣ που δείχνουν την αλληλευτική προσπάθεια, δηλαδή ώρα αλίας ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, στο, στην υφαλοκρηπίδα, κάτω πέρα από τα 200 μέτρα, βλέπετε ότι στα κάτω από 200 μέτρα και στα 200-500 είναι ψηλά από τα 800 και πάνω η αλληλευτική προσπάθεια είναι χαμηλή. Δηλαδή, η αλληλεία ε, του Γρεναδιέρου και της Μουρούνας είναι κάτι που γίνεται κυρίως ψηλότερα στην υφαλοκρηπίδα και όχι στα πολύ χαμηλά. Το δεξί τώρα, ε, η δεξί, το δεξί γράφημα είναι της Γαλλίας, δείχνει την αύξηση της ελευτικής προσπάθειας σε βαθιά νερά, πέρα από τα 800 το λέμε αυτή τη στιγμή, από το 2003 και μετά. Εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που ξεκίνησε από το 2003 και μετά, που μείωσε την προσπάθεια ή όπου οι στολίσκοι προσαρμόστηκαν στις νέες εξελίξεις. Η τελευταία τώρα είναι ώρε, η τελευταίο, το τελευταίο γράφημα είναι ώρες αλίευσης και επιφάνειες, παρόμοια στοιχεία βλέπουμε, για τα Ιρλανδικά ύδατα. Εδώ βλέπετε τώρα μία ε, χωρική κατανομή της αλλιευτικής προσπάθειας. Στο δεξί γράφημα βλέπετε στην Ιρλανδική θάλασσα τη μείωση του χρόνου ανα, ε, και στα ύδατα της Βρετανίας την κατανομή όλων των ειδών αλίευσης σε βαθιά νερά. Βλέπετε ότι η, προσπά, η αλευτική προσπάθεια των σχετικών των σκαφών γίνεται κατά βάση στα χωρικά ύδατα, στην υφαλοκρηπίδα. Τώρα, από ένα άλλο παράδειγμα από τον ε, κόλπο της ε, Βισκάια, το Βισκαϊκό κόλπο στην, ε, στον Ατλαντικό που αυτή τη στιγμή βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ε, εκφόρτωσης ψαριών από του βαθιού νερού, ωστόσο η μελέτη έγινε για αλίευση όχι βαθιών, υδάτων και όπου δεν εφαρμόζονται δεν έχουμε λάβει υπόψη τη τροποποίηση του κανονισμού. Έχουν γίνει πολύ περισσότερε μελέτε προφανώς στα ευάλωτα ε, οικοσύστηματα VME στην, ε, στο, στο πλαίσιο του Coral Fish και στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Weaver. Τώρα, επιπτώσεις διαχείρισης. Οι αλληλευτικές προσπάθειες στα βαθιά νερά μπορεί να εκτιμηθούν με ακριβή χρησιμοποιότητα στοιχεία παρακολούθηση των σκαφών με δορυφόρο, το VMS. Αυτό καλύπτει όλα τα σκάφη, αν και υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα. Η ρύθμιση της αλληλείας e αυτής ήταν αποτελεσματική για τη μείωση της, αλληλευτικής, της υπερβολικής αλληλευτικής προσπάθειας. Αυτό το είπα, αναφέρθηκε ήδη. Τώρα, το, το εδαφικό ίχνος της Αλίας e μειώθηκε μετά το 2000. Η ελευτική προσπάθεια στο άνω τμήμα της ε, αλλιεύσης που αλλιεύουν μερλούκιο, βατραχόψερο η ε, μαύρη πολλάκα είναι πολύ ψηλότερα από τις προσπάθειες που γίνονται στα βαθύτερα νερά. Ο αντίκτυπος στα, οικολογικά, στα ευάλωτα οικολογικά συστήματα δεν δημιουργείται μόνο από την αλίευση σε βαθιά νερά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ε, ως εκ τούτου χρειάζεται να υπάρξει μια προσέγγιση χωρικής διαχείρισης που δεν περιορίζεται μόνο στα είδη βαθέων υδάτων, αλλά συνολικά. Να σας δώσω τώρα δύο στοιχεία για τον τρόπο αξιολόγηση των αποθεμάτων, αν και περιλαμβάνεται και στη νέα έκθεση, αξιολόγηση των αποθεμάτων. Σε πολλά ήδη τα στοιχεία είναι data που δηλαδή χωρίς ε, ανεπαρκή, ιδίως τώρα ωστόσο με βάση στοιχεία που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορούμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία και μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση περισσότερα. Εδώ δεξιά βλέπετε σε κόκκινο τις μελέτες περιπτώσεων όπου το Deep Fishman έδωσε νέες μεθόδους αξιολόγησης των αποθεμάτων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα για τις μεθόδους αξιολόγησης που εξετάζουμε. Απλά να σας πω ότι η αξιολόγηση δημιουργούνται κατηγορίες αξιολόγησης, κάποιες στηρίζονται σε τάσεις, κάποιες σε δείκτες, έχουν, υπάρχουν και δείκτες και τέλος γίνεται αξιολόγηση στρατηγικής διαχείρισης. Η, σε ό,τι αφορά το τη μουρούνα, την μπλε μουρούνα, το είπε ο κύριος είναι κάτι που το αναπτύξαμε γιατί ένα από τα μοντέλα αξιολόγησης της μπλε έγινε στα πλαίσια του, Deep Fishman. Εδώ έχετε μια διαφορετική αξιολόγηση για τον ε, Γρεναδιέρο που ωστόσο για τον οποίο ωστόσο αντιμετωπίζουμε προβλήματα γιατί είναι συχνό bycatch. Είναι μια... Ακολουθούμε λοιπόν μια ημιποσοτικοποιημένη ανάλυση που έχει τη δυνατότητα να δούμε τον αντίκτυπο που έχει στο καθρεπτόψαρο αυτή η παρεπόμενη αλίευση από το 2006 και μετά. Συμπεράσματα τώρα, νομίζω ότι... Τι να σας τα πω, σας τα είπα και θα πάω κατευθείαν στις υφιστάμενες δραστηριότητες, στις υφιστάμενες εργασίες, στις συνεχιζόμενες εργασίες. Είδαμε, προσπαθούμε να δούμε τον αντίκτυπο στον πυθμένα, κάτι που χρειάζεται περαιτέρω με, μελέτη. Θα δουλέψουμε στα πλαίσια του Deep Fish με ένα άλλο έργο που λέγεται Coral Fish, δεν θα σας τα παρουσιάσω εδώ σήμερα, αλλά χρειάζονται Χρειαζόμαστε μια βάση δεδομένου για τα ευάλωτα θαλάσσια ενάλλια οικοσυστήματα και την χωρική διαχείριση των ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση, βάση δεδομένα της ΦΑΟ. Επίσης θα προχωρήσουμε να κάνουμε μια σειρά σεναρίων προσωμείωσης ε, διαχείρισης είδος και αναμέγεθος και εργασίες για το trade-off, ε, τον συμβιβασμό μεταξύ συντήρησης και διαχείρισης. Κάθε μορφής, κάθε διαχείριση ανθρώπινη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το trade-off. Το ερώτημα είναι πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς ένα χ είδος χωρίς να έχεις υπερβολική εθνισμότητα του είδους και αρνητικές επιπτώσεις στα ευαίσθητα βαθέα οικοσυστήματα. Τώρα, για τους ε, καρχαρίες δεν έχει ολοκληρωθεί το, η μελέτη, αλλά προσπαθούμε να δούμε αξιολόγηση των ε, ε, σκυλοψάρων αυτών. Συνεχίζεται η συζήτηση. Πάντως, τώρα, ο αντίκτυπος. Αυτό είναι μια αμφιλεγόμενη συζήτηση. Σας έδωσε ένα παράδειγμα μιας μελέτης που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Ερμιώνη στη Μεσόγειο που δείχνει ότι η αλία, η γαριδών σε βαθιά θάλασσα στην Μεσόγειο έχει τρομερά αρνητικές συνέπειες. Τώρα, 15.000 τόνους το χρόνο είναι οι γαρίδες στη Μεσόγειο και τι σημαίνει αν δεν βρούμε στην ευρωπαϊκή αγορά 15.000 τόνους γαρίδες. Κάτι άλλο, ίσως γαρίδες από τα τοπικά νερά ή σε υδατοκαλλιέργεια, κάτι που γίνεται σε δομές που δημιουργούνται δι, αντί για μαγκρόβιες, κάτι που είναι εξαιρετικά ε, προβληματικό και δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Σακάου Σακάου-Κουαδράδο. Ε, Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Από το 2004 οι συζητήσει για τα ευάλωτα θαλάσσια οικοσύστηματα λαμβάνουν χώρα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτή η διαδικασία το 2006 κορυφώθηκε με την ε, υιοθέτηση του ψηφίσματος 61 του 2005 που ε, καλή της ε, πόδα να προσδιορίσουν τα βάλωτα ε, ε, θαλάσσια οικοσυστήματα και να τα προστατέψουν από τις αλληλευτικές δραστηριότητες βυθού. Υπό το φως αυτού του ψηφίσματος και ως απαραίτητο βήμα για τον προσδιορισμό αυτών των ευάλωτων οικοσυστημάτων, η Ισπανία από μόνη της σε συνεργασία με άλλα κράτη από το 2005 και μετά ξεκίνησε ένα δαπανηρό και φιλόδοξο πρόγραμμα χαρτογράφησης του βυθού σε διάφορα σημεία του ωκεανού. Ως ε, παραδείγματα έχουμε ε, διάφορα ε, project από το 2005 μέχρι το 2008 για παράδειγμα ένα πρόγραμμα ένα άλλο το Atlantis από το 2007 μέχρι 2010 με επιφάνεια 59.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων στην Παταγωνία. Ένα άλλο project, το Rapsur, από το 2008 στο 2010 με 16 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αλλά εγώ εδώ θα σας ε, θα περιοριστώ στο πρόγραμμα Νερέιτα στην περιοχή του Νάφο. Το ψήφισμα 66 που υιοθετήθηκε το 2011 αναγνώριζε την ανάγκη προγραμμάτων χαρτογράφησης για να εντοπιστούν αυτά τα ευάλωτα οικοσυστήματα. Το πρόγραμμα Νερέιδα είναι ένα πολυεπιστημονικό project με συμμετοχή διαφόρων φορέων από τον Καναδά, τρία ε, Ινστιτούτα του Καναδά, Στη Ρωσία, που έχουμε το Ινστιτούτο Σίρσοφ, από το Ηνωμένο Βασίλειο το ΣΕΦΑΣ και βέβαια από την Ισπανία, που έχουμε το Κοινοβακικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θαλασσών. Ο γενικός ε, στόχος του σχεδίου αυτού ήταν η εφαρμογή ε, της προσέγγισης οικοσυστήματος ε, στην διαχείριση της αλληλευτικής προσπάθειας για να προστατευτούν αυτά τα ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα ιδιαίτερως τα είδη των σφουγγαριών και των κοραλιών ε, ψυχρών υδάτων. Η ειδική στόχη είναι να εντοπιστούν οι, ε, να εντοπιστούν οι οργανισμοί που ε, συμμετέχουν σε τέτοιου οικοσυστήματα, να περιγραφεί η οικολογία των ε, βαθέων, των οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων, να γίνει χαρτογράφηση αυτών και να, να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ένα σύστημα, μια βάση δεδομένων με όλες τις πληροφορίες που θα ε, συλλεγόντουσαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού. Οι έρευνες ε, του Νερέιδα έλαβαν χώρα από το, τα έτη 2009 και 2010 με δύο ερευνητικά σκάφη. Αριστερά έχουμε το ισπανικό ε, σκάφος Μιγγέλ Όλιβερ και δεξιά έχουμε το Χάτσον που είναι καναδέζικο ερευνητικό σκάφος. Πάνω σε αυτά τα σκάφη είχαμε ε, ε, επιστήμονες διαφόρων δικοτήτων, χαρτογράφους, οικολόγους, υδρογράφους κλπ. Η περιοχή καλύπτει αυτή μια περιοχή ανάμεσα ε, στα 700 και τα 2.000 μέτρα βάθους ανοιχτά στον βορειοδυτικό Ατλαντικό ωκεανό. Ε, έξι συνολικά πολυεπιστημονικές έρευνες ε, έγιναν τα έτη 2009 και 2010 στο από το Μίγκελ Όλιβερ και επιπλέον το καναδικό σκάφος, του Χάτσον, ε, διενήργησε δύο οπτικές έρευνες που ε, κάλυψαν μια περιοχή 69.000 περίπου τετραγωνικών χιλιόμετρων. Συλλέχθησαν διαφόρων ειδών στοιχεία ε, υδρογραφία για παράδειγμα, υδρογραφικά στοιχεία μέσω CTD, είναι μια διάταξη που ε, μας δίδει πληροφορίες για ε, τις στήλες ύδατος, περιεκτικότητα σε άλλα, θερμοκρασία κλπ. Και βάθος. Ένα άλλο τμήμα του project αφορούσε τη χαρτογραφία, χαρτογράφηση για την ακρίβεια, ε, η χαρτογράφηση έγινε ε, από το Μιγέλ Όλιβερ με ένα ηχοβολιστικό μηχάνημα πολλαπλής δέσμης που μας δίνει μια πλατιά εικόνα του βυθού με πληροφορίες για την μορφολογία του, ε, τις χαράδρες και οποιασδήποτε άλλες δομές μπορεί να βρούμε στο βυθό. Συνολική ε, περιοχή που καλύφθηκε είναι περίπου 69.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επιπλέον, πήραμε πληροφορίες από, υποπεριοχή, από ε, μέσω bottom profilers, ε, το συγκεκριμένο μηχάνημα ονομάζεται TOPAS, που μας δίνουν πληροφορίες για ε, βάθος κάτω από το βυθό. 30, ε, μέχρι 30 εκατοστά μέσα στο βυθό. Οι γεωλογικές πληροφορίες από την άλλη μεριά εντοπίσαμε 13 διαφορετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά για τα οποία πήραν πληροφορίες, ε, χαράδρες, ε, ζήματα οι περιοχές ζημάτων δηλαδή κλπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας ε, δίνουν μια περίληψη ε, του γεωλογικού προφίλ ε, της περιοχής για να τις να πληροφορίες τις οποίες συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε. Ε, τα ερευνητικά σκάφη ε, ήταν εξοπλισμένα ε, με διατάξεις και εξοπλισμό που επέτρεπαν τη μελέτη του βυθού. Αφενός είχαμε, τις, είχαμε δράγες, βυθοκόρους δηλαδή κατά βάση, που για σκληρούς πυθμένες μας δίνουν πληροφορίες για τον τύπο του ε, πετρώματος ή του υλικού ε, καθώς επίσης και για τα ζώα, τα οποία, τους οργανισμούς μάλλον που ζουν ε, σε αυτούς τους βυθούς. Για τους μαλακούς βυθούς χρησιμοποίησαμε τον box scorer, που μας δίνουν ένα κύβο ε, ειζήματος αντιπροσωπευτικού για την περιοχή την οποία ερευνούμε. Ένα άλλο τμήμα του project ήταν η χρήση βίντεο, βιντεοσκόπησης, και φωτογραφικών μηχανών υψηλή ευκρίνειας και που μας έδιναν εγκάρσιες τομές. Ε, προσπαθώ εδώ να σας δώσω μια σύνοψη των σημείων ε, τα οποία επιλέξαμε ως δείγματα, ε, τα μικρά διαμαντάκια που βλέπετε εδώ, 105 ε, δείγματα συγκεκριμένα ε, με τη Δράγα. Ε, με το box scorer ε, το ίδιο, αλλά είχαμε διαφορετικά σημεία, 368 δείγματα συγκεκριμένα με το box scorer. Εδώ βλέπουμε δύο εγκάρσιες τομές, τις, τις οποίες έβγαλε το Hudson Η περιοχή αυτή τώρα είναι κλειστή για την αλίευση, απαγορεύεται η αλίευση. Ε, υπάρχουν πολλά σφουγγάρια, βλέπετε, ε, λιβάδια από σφουγγάρια. Πάνω από 2.000 φωτογραφίες και 116 ώρες βίντεο ελήφθησαν από το καναδικό σκάφος. Βλέπετε μερικά δείγματα εδώ. Σε αυτή τη διαφάνεια προσπαθώ να δώσω μια σύνοψη, μια περίληψη ορισμένων των, από τις δράσεις και ε, τις αποφάσεις που ο ΝΑΦΟ πήρε για να προστατεύσει αυτά τα ευάλωτα θαλάσσια αποστήματα. Το 2007 συγκεκριμένα τέσσερις, τέσσερα θαλάσσια όροι ε, έκλεισαν για την ε, Αλία Βυθού. Το 2008 δημιουργήθηκε μια ζώνη προστασίας κοραλιών στην περιοχή 3 όμικρον. Το 2009 έκλεισαν δύο ακόμα θαλάσσια όροι. Το 2010 11 περιοχές έκλεισαν για την Αλία Βυθού για να προστατευθούν κοράλια και σφουγγάρια. Ο χάρτης που έχουμε με τις ε, ε, πραγματικές περιοχές που έχουν κλείσει είναι αυτό, 18 συγκεκριμένα ε, περιοχές του ΝΑΦΟ είναι κλειστές, τη χάνουν σε απαγόρευση αλίευση βυθού. Η σημερινή κατάσταση στην περιοχή που διανοήθηκε τον Ερέιδα έχει 11 περιοχές τις οποίες εντοπίσαμε για μέσω των ερευνών για βαθύβια ψάρια και έχουν κλείσει προκειμένου να προστατευθούν τα κοράλια και τα σουγκάρια. Αυτές οι 11 περιοχές που έχουν κλείσει ε, αντιπροσωπεύουν περίπου 8.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Με όλες αυτές τις ε, πληροφορίες των ερευνών μας ε, είναι, δύο, δύο οδηγοί, ε, ένας για κοράλια και ένας για σφουγγάρια από τον άφο. Ε, αυτές οι περιοχές ε, μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ακριβείς με βάση τις πληροφορίες που λάβαμε από το, από το πρόγραμμα Νερέιδα. Η, η, η Επιτροπή ε, αλίας το 2014 θα ξαναδεί τα στοιχεία και ενδεχομένως θα αλλάξει τις περιοχές. Τα... Ε, ε, εμείς χρειάστηκε να καθορίσουμε κάποιες προτεραιότητες για τη μελέτη των κλειστών περιοχών. Εδώ βλέπουμε ένα πίνακα που δείχνει πόσα δείγματα λάβαμε για κάθε μία από αυτές τις κλειστές περιοχές. Ε, καθόρισαν προτεραιότητες λοιπόν, ψηλέ και χαμηλότερες προτεραιότητες για την μελέτη κάθε μιας από αυτές τις κλειστές περιοχές. Σήμερα δύο κλειστές περιοχές έχουν μελεθεί πλήρως, η έξι, το Sackville Spur, και τα αποτέλεσματα της ανάλυσης παρουσιάστηκαν στην ομάδα εργασία του ΝΑΦΟ για την προσέγγιση κατά υποσυστήματα στη διαχείριση αλίας και δεν άλλαξε ο χαρακτηρισμός, παρέμεινε κλειστή περιοχή. Η άλλη περιοχή που μελετήθηκε ήταν η παρθμόν 5, η Flemish ε, Pass Eastern Canyon ε, και η, τα, ε, τα μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει η οριογραμμή να διευρυνθεί στα 2.500. Η δηλαδή θα μπορεί στην περιοχή θα πρέπει να διευθύνει στα, σε βάθος 2.500 μέτρων. Η αναθεώρηση των κλειστών περιοχών θα γίνει το 2014 από την Επιτροπή Αλίας. όπως σας είπα. Οπότε οι μελλοντικές δραστηριότητες του Νερέιδα θα εστιαστούν στο να κάνουμε ανάλυση βίντεο του Flemish Cup και των κλειστών περιοχών για να αξιολογήσουμε, να πάρουμε πληροφορίες σχετικά μάλλον με την αξιολόγηση της βιοπικιλότητας σε σχέση με, τα, με τους οργανισμούς που ζουν εκεί. Θέλουμε μια πλήρη ανάλυση των δειγμάτων της δράγας. Ε, θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση των δειγμάτων του Box Scorer γιατί μας δίνουν μια ποσοτική περιγραφή των μαλακών βυθών. Ε, μόνο 40 από 468 δείγματα έχουμε επεξεργαστεί αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την επεξεργασία και πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι αναλύσεις είναι κρίσιμες για την αναθεώρηση ε, των κλειστών περιοχών του ΝΑΦΟ γιατί είναι η μόνη πηγή ε, στοιχείων για, τις, ε, για τα βαθαία ύδατα που υπάρχουν και καλύπτει τις κλειστές περιοχές του ΝΑΦΟ. Τώρα, το κατά πόσο θα διευρυθεί και θα επεκταθεί αυτή η δραστηριότητά μας, αυτό μας το project, θα εξελθεί από τη χρηματοδότηση. Αυτά ήθελα να σα πω για το project μα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σακάου. Ε, όπως συμφωνήσαμε στην Επιτροπή, ε, θα Έχουμε τρεις ε, προσκαλισμένους και θέλω να τους δώσω το λόγο όχι ως εισηγητές, ε, αλλά για να τοποθετηθούν τρία-τέσσερα λεπτά ο καθένας. Ε, ο πρώτος τώρα και οι δύο υπόλοιποι στο, μετά το τρίτο πάνελ. Λοιπόν, θα δώσω λοιπόν, το λόγο στον πρώτο προσκαλισμένο μας, την πρώτη προσκαλισμένη, την κυρία Σουασίκ Λεγκάλ. Παρακαλώ. Λουγκάλ. Λουγκάλ για την ακρίβεια. Euh, Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο που δίνει το λόγο σε μια επαγγελματία της Αλίας. Είμαι ε, ε, από την ε, Φινιστέρ της Βρετάνης. Ε, είμαι διευθύντρια ε, ε, ενός ε, ε αλληλευτικού ε, στόλου, 11 συγκεκριμένες, συγκεκριμένα τράτες, 24 μέτρων, 24, συγγνώμη, 80 στη θάλασσα και 17 στη στεριά, ε, αλής και προσωπικό, 3.700 τόνοι αλλιευμάτων αναχρόνου το ε, ε, ε, συγγνώμη, έχω λίγο τράκ γιατί δεν έχω συνηθίσει να μιλάω σε κοινό. Ε, υπάρχουν και μικρά σκάφη λοιπόν που αλλιεύουν σε μεγάλα βάθη. από τα 120 έως τα 800 μέτρα συγκεκριμένα εμείς. Ε, εμείς ε, κυρίως αλλιεύουμε πεσκαντρίτσα. Ε, το 10% των ειδών που αλλιεύουμε ε, είναι βαθύβια είδη. Σπαθόψαρο, ε, ε και ε, Μουρούνα. Ε, υπάρχουν όμως και άλλα σκάφη τα οποία δεν έχουν άδεια ε, για αλλή βαθέων υδάτων αλλά ψαρεύουν στα 400 850 μέτρα και απορρίπτουν τα λίγα ε, αλλιεύματα βυθού βαθιών υδάτων που πιάνουν. Επομένω και αυτοί επηρεάζονται από τα μέτρα που συζητούμε. Επίσης ήθελα να σας πω ότι μιλήσαμε για κοράλια οι αλληλείς μας είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένοι και δεν έχουν κανένα συμφέρον να αλλιεύουν κοράλια, γνωρίζουν τις ζώνες των κοραλιών. Τα κοράλια πραγματικά μας δυσκολεύουν, διότι καταστρέφουν τις στράτες, τα δίχτυα μας. Συνεπώς δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε να αλλιεύσουμε σε ζώνες με κοράλια. η αλήθεια είναι σχετικά έξυπνοι άνθρωποι. τα σκυλόψαρα, ούτε τα σκυλόψαρα ε, μας αρέσουν, γιατί επίσης τα σκυλόψαρα ε, ε, με το δέρμα τους ε, τρώνε τα ψάρια τα οποία έχουμε ήδη πιάσει. Συνεπώς οι πελαγίες αποφεύγουν και τις ζώνες με σκυλόψαρα. Του λεχθέντος, δεν σας είπα πού ψαρεύουμε. Ψαρεύουμε από το νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας μέχρι τον 406ο παράλληλο περίπου. Γνωρίζουμε πολύ καλά, οι αλλιές μας γνωρίζουν πολύ καλά αυτή την περιοχή και ε, προσπαθούν ε, να αλλιεύουν με τρόπο βιώσιμο. Μάλιστα, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, βλέπουν μια πραγματική αύξηση των ε, αλλιευμάτων ε, συγκεκριμένων ειδών τουλάχιστον, όχι όλων, όπως για παράδειγμα του σπαθόψαρου. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στα μέλη μας. Τρεις έχουν ζητήσει το λόγο. Κυρία Τόμας. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς τον κύριο Λοραντς που μας είπε ότι στην απαγόρευση, για παράδειγμα, του ε, σπαθόψαρου που οδηγηθήκαμε σε αύξηση, του καθεπτόψαρου, συγγνώμη, αυτόν οδηγηθήκαμε σε αύξηση των παρεπόμενων ειδών. Είπατε επίσης ότι η χωρική διαχείριση είναι μια λύση. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερο πράγματα για αυτή τη δημιουργία ζωνών ε, στους πυθμένες. Και μία ερώτηση και προς την κυρία Μαρσακάου Κουαδράδο. Προφανώς όλοι οι πυθμένες δεν έχουν, δεν είναι κοραλογενείς, ούτε είναι και ευάλωτοι. Οι μελέτες που έχετε κάνει και οι ζώνες απαγόρευσης αλίες οδηγούν και αυτές την ε, απαγόρευση αλίας και κλείσιμο περιχάραξη συγκεκριμένων ζωνών. Αν ναι, ε, η απάντηση είναι ότι όλα πηγαίνουν προς τη δημιουργία ζωνών. Σωστά τα καταλαβαίνω. Ευχαριστώ κυρία Τόνα μας. Ή δεν κατάλαβα καλά, ή τέλος πάντων διευκρινίστε μου κάτι. Δεν είπα ότι θα μιλήσει μόνο όποιος δεν μίλησε στον πρώτο γύρο. Θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους πρώτα και μετά σε εσά. Ο κύριος Πέλμο Μωράτο. Τέσσερα-πέντε λεπτά. Καλησπέρα σας. Ε, εγώ είμαι ερευνητής ε, βιολόγος ε, που ασχολείται με θέματα ηλίας, Πορτογάλος. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια ήταν το να συνδέσουμε κάπως ε, τα διάφορα ε, αλληλευτικά εργαλεία έτσι ώστε να συγκρίνουμε και τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. Και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Να σας δώσω έτσι μία πληροφορία για να σχηματίσετε κι εσείς μια άποψη. Ας δούμε λιγάκι μία ε, περίπτωση μελέτης ε, το πράξαμε αυτό και καταλήξαμε στο ότι Μία ε, μηχανότρατα βυθού είναι σαν να χρησιμοποιείται 16 μέχρι 25.000 απλάδια. Έτσι λοιπόν, Το ίδιο ισχύει και στην χρονική προέκταση. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κατά κάποιον τρόπο πώς, ε, ποιες είναι οι διαφορετικές επιπτώσεις, πώς ποικίλουν επιπτώσεις από τη χρήση διαφόρων εργαλείων, αλληλευτικών εργαλείων. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχουν και εναλλακτικέ λύσεις. Ε, μπορούμε να συνεχίσουμε την αλία, ίσως ε, περιορισμένη βέβαια, με μικρότερες επιπτώσεις. Ακόμα και αν ε, συγκρίνουμε τα πλάδια με τις ε, τράτες, ε, τα απλάδια βοηθούν στο να καλύψουμε τα παραγάδια, βοηθούν να Έχουμε αλληλεία με απασχόληση και σε ορισμένε περιπτώσεις έχουν και οικονομική αξία. Γιατί και η ποιότητα των ψαριών που πιάνονται με παραγάδια είναι πολύ καλύτερη. Άρα δηλαδή υπάρχει ελπίδα και όσον αφορά τα ε, ψάρια βαθέως βιτού, ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις, ποιες μπορούν να χρησιμοποιηθούν που να προκαλούν μικρότερη ζημιά στο οικοσύστημα. Ευχαριστούμε και για την παρέμβαση και για την ε, σαφήνεια και λιτότητα των παρεμβάσεων. Ο κύριο Βότλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Νομίζω ότι εδώ το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να δούμε λιγάκι το ότι δεν πρόκειται εδώ μόνο για τα ψάρια, αλλά πρόκειται γενικά για την καταστρεπτικότητα, την καταστροφή που προκαρούν οι τράτες βυθού στο οικοσύστημα. Αναζητήσαμε ε, στοιχεία στην επιστημονική λογοτεχνία, βιβλιογραφία και είδαμε ότι υπάρχουν 74 μελέτες που καταδεικνύουν ότι με τη χρήση μηχανότρατας βυθού ε, προκαλούνται μεγάλες μιας καμία μελέτη δεν λέει ότι είναι καλή αυτή η τράτα. Ε, προκαλεί μεγάλη ζημιά και επίσης όλες οι μελέτες ισχυρίζονται ότι οι ζημιές προκαλούνται όχι μόνο στο βορειοατλαντικό αλλά και στο Νότιο Ειρηνικό, στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία και εκεί προκαλούνται μεγάλες ζημιές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί κανείς να ισχυριστεί το ότι ε, δεν είναι σίγουρο ή είναι αμφίβολο κατά πόσον οι μηχανότρατες ε, βυθού προκαλούν ζημιά ή όχι. Επίσης, ε, όσον αφορά τα ψάρια βαθέως βυθού. Αυτά που λέγονται για τα ψάρια βυθού ισχύουν και για αυτά που ζουν σε βάθος 800 μέτρων. Για τα περισσότερα είδη χρειάζεται μία ικανοποιητική περίοδος ανασύστασης. Εγώ είμαι ε, βιολόγος και ασχολούμαι κυρίως με τα αγκαθωτά κοράλια. Σε γενικές γραμμές τα αγκαθωτά κοράλια ε, ζουν το ελάχιστο 50 χρόνια και κατά το μέγιστο 100 χρόνια. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα να ανασυσταθεί αυτό το είδος ε, ε, βαθέως βυθού είναι πάρα πολύ μικρές. Η γυναίκα μου, ή η κόρη μου θα έχει πια γεράσει όταν θα υπάρξει ανασύσταση αυτού του είδους και ίσως να γεράσει και η κόρη της. Μιλάμε για τέτοιου είδους χρονικά διαστήματα. Επίσης πιστεύω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δυστυχώς αυτά δεν μπορεί κανείς να τα δει. Εγώ ε, είμαι πολύ τυχερός, ε, έκανα πάρα πολλές καταδύσεις και ξέρω ε, ποια είναι η εικόνα αυτών των ειδών του βαθέως βητού. Εάν όμως μιλάγαμε για άλλα είδη τα οποία βλέπουμε, εκεί θα υπήρχε οργή στο κοινό και θα γινόντουσαν πάρα πολλές συζητήσεις. Εδώ λοιπόν ε, πρέπει να προσέξουμε ε, το ότι δεν βλέπει κανείς κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν απαγορεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, περνάμε με την κυρία, κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο συνεχίζει η κυρία Πατραωνέβης. Ωραία. Η ερώτησή μου αφορά την κυρία Μαρ Κουαδράδο. Νομίζω ότι κατέτσι πως μέσω μιας καλής επιστημονικής έρευνας είναι δυνατόν να εντοπίσουμε και να ε, καθορίσουμε τα πιο ευάλωτα οικοσυστήματα, θαλάσσια οικοσυστήματα, τα οποία θα, ε, στα οποία θα πρέπει να απαγορεύεται η αλήψη με συγκεκριμένα εργαλεία, με συγκεκριμένες μεθόδους, αυτές τις μεθόδους δηλαδή που έχουν τις πιο αρνητικές συνέπειες. Ε, αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε να επενδύσουμε στην επιστημονική έρευνα για να εντοπίσουμε αυτές ακριβώς τις περιοχές. Η ερώτησή μου είναι εξή. Πώς, ε, μάλλον, τι κόστος είχε, είχαν αυτά τα project. Τελειώσατε την ε, παρουσίασή σας λέγοντας ότι χρειάζεται και άλλη χρηματοδότηση για να συνεχίσετε. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω ε, γιατί ποσά μιλούμε ακριβώς, ε, για ποιο χρονικό διάστημα και πώ ακριβώς εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ως τώρα. Φράγα. Κυρία Φράγα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν μια σκέψη σε σχέση με την, ε, με την Deep Fishman. Θα ήθελα να πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πλήρωσε, μάλλον ζήτησε και πλήρωσε αυτό το μεγάλο project. Τρία εκατομμύρια ευρώ ήταν το κόστος του Deep Fishman. Αυτό που με εντυπωσιαζεί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τελειώσει αυτό το project υπέβαλε πρόταση. Δηλαδή <laughs> υποβλήθηκαν προσωρινά συμπεράσματα, αλλά ακόμα το project δεν έχει καν τελειώσει. Οπότε η ερώτηση αυτή απευθύνεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς είναι δυνατόν να ε, παραγγέλει, να χρηματοδοτεί ένα τόσο σημαντικό project και πριν γίνουν γνωστά τα πορίσματα υποβάλλει προτάσεις που ούτε καν βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση με τα προσωρινά συμπεράσματα. Θα ήθελα να κάνω και την εξή ερώτηση. Μεταξύ των προτάσεων που κάνετε για βαθύ είδη, σε σχέση με τα παρατήματα 1 και 2 που στην καινούργια πρόταση ενοποιούνται, ε, κάνετε κάποιες συστάσεις τις οποίες εν μέρη δέχτηκε η Κομισιόν, εν μέρη όχι. Προτείνατε για παράδειγμα ε, τι να ληφθούν υπόψη οι κατάλληλοι του ΝΕΑΦ. Ποια είναι η άποψή σας είχατε πει να συμπεριληφθούν και άλλα είδη τα οποία δεν συμπεριλήφθησαν. Για παράδειγμα το σκορπίδι. Ε, ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν για αυτή την ε, ε, μονομερική αποδοχή των ε, ειδών που προτείνεται. Δεύτερον, ερώτηση προς την κυρία Σακάου μίλησε για το project του ΝΑΦΟ. θα μπορούσατε να μας μιλήσετε και για το project της ζώνη ΝΑΦ και αν έχετε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Τρίτον, σχόλιο και ερώτηση. Τι παράξενο όλα τα μεγάλα project που λαμβάνουν χώρα ε, χρηματοδοτούμενα είτε από την, την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τα κράτη-μέλη είτε από διεθνείς ε, οργανισμούς όλα κινούνται στην γραμμή των ΗΕ, Εθνών, δηλαδή ε, της προσέγγισης σαν οικοσύστημα. Ακολουθούν δηλαδή τις συστάσεις του ΦΑΟ και των ΗΕ. Εθνών. Πώς είναι δυνατόν όλες οι εκθέσεις, όλες οι μελέτες να βαίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και η πρόταση Κομισιόν να απορρίπτει ο, αυτήν ακριβώς την προσέγγιση, όλα αυτά τα project, όλα αυτά τα πορίσματα και να υπαγορεύει την απαγόρευση. Τέλος, η πλήρης απαγόρευση της ε, χρήσης ε, ε τράτας βυθού. Τι, συμπερα... αποτελέσματα θα έχει. Ε, μήπως ε, θα αυξήσει τον αριθμό των σκυλόψερων, ας πούμε, κάτι που είναι κακό. Και η, η απαγόρευση αυτή, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ε, συμφωνώ με την κυρία Τόμας. Ή, για ενδεχομένως μια προσέγγιση αναζώνες θα ήταν πιο, το πιο κατάλληλο μέτρο. Γιατί προς τα εκεί μας οδηγούν οι έρευνες. Η Κομισιόν πρέπει να μας εξηγήσει γιατί πάντοτε πρέπει να κινείται αντίθετα με το ρεύμα αντίθετα με τα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή σε διεθνέ και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριο Σκάντεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια παρατήρηση προς, τον, προς την Πορτογαλίδα επιστήμονα φίλη μας. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο εύκολα περνάει. Μας έλεγε ότι το παραγάδι που είναι ε, που είναι ε, αλλιευτικό εργαλείο ε, έχει μεγαλύτερη επίπτωση από ότι το, ε, το απλά ε, δεν έχει νόημα όταν το ένα έχει 600 χρόνια ιστορία και το άλλο μικρότερη. παρατήρηση. Προς την Επιτροπή θέλω να θέσω μια ερώτηση. Όπως και η κυρία φράγκα χοντρικά. Γιατί δεν περιμένετε τα αποτελέσματα τα οριστικά, τέλο πάντων οριστικά δεν είναι ποτέ, αλλά τα τελικά αποτελέσματα του Deep Fishman που στήχησε κάμποσα φράγκα πριν ε, υποβάλλετε την πρότασή σα. Δεν στέκει. Θα μπορούσατε να περιμένετε. Λίγοι μήνες ακόμα μένα για να τελειώσει η μελέτη και θα είχατε με τα κειμενικά στοιχεία. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν, γιατί το κάνατε. Και επιπλέον, πρέπει να έχουμε χρόνο για να μιλήσουν όλοι. Όπως και οι κυρίες Φράγκα και το ΜΑ, πιστεύω και εγώ ότι η αρχή της δημιουργία ζωνών είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πρώτο, παγώνουμε το αποτύπωμα. Δεύτερον, δημιουργούμε ζώνες. Κάτι θετικό και ενδιαφέρον. Ο κ. Αρσένης. Thank you very much, Chair. I also... Κοιτάξτε και εγώ ε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε ο καθηγητής από την Πορτογαλία, ο κ. Μωράτος. Δηλαδή, ένας χρόνος χρήσης Μηχανότρωτας σημαίνει μέχρι και 600 χρόνια χρήση παραγαδιών. Και θα ήθελα να ρωτήσω ε, τους ε, δύο προσκεκλημένους μας αν μπορούν να σχολιάσουν αυτήν την, αυτόν τον ισχυρισμό. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω και τον κύριο Λεωρόν στο εξής. Μας είπαν ότι ο βασικότερος στόχος του project Deep Fishman ήταν να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι μέγιστες ελεύσιμες ποσοστώσεις, τα TAC, και όχι τόσο να ερευνηθούν ε, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή η ε, έμφαση αποδίδεται στα TAC και όχι τόσο στα λεπτικα εργαλεία. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Αρσένη. Οι δύο εισηγητές έχουν το λόγο για να δούμε όπως θέλετε με τη σειρά. Πρώτη κύριε Σακάου, ο κύριος Βεράνς. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο. Adelante. Venga. Ο κύριος Λοράνς. προτείνω όπως και οι προηγούμενοι, οι αμβολητές στο προηγούμενο πάνελ. Για την ερώτηση της κυρίας Η μείωση της πίεσης στα, ήδη, στα βαθύβια ήδη, έχει επιπτώσεις και στα άλλα, ναι. Είναι ένα γενικό φαινόμενο σε, όλες τις μορφές, σε όλα τα ίδια ελίματα. Η βιβλιογραφία για τα ίδια αυτά έλεγε, μιλούσε για υπερεκμετάλλευση που έχει αρνητικές επιπτώσεις και στα βαθύ είδη και στο οικοσυστήματα. Ο στόχος ήταν να υπάρχει ένα ε, σοβαρό, ένα, ένα κανονικό επίπεδο για τα εμπορικά είδη και αυτό έχει επιπτώσεις άμεσα και στα υπόλοιπα. Όταν βελτιώνουμε την κατάσταση για τα εμπορικά είδη, βελτιώνουμε και τα υπόλοιπα. Για τη δεύτερη ερώτηση της κυρίας Τωμά χωρική διαχείριση είναι λύση. Δεν θα μιλήσω για το πρόγραμμα Coral Fish που δεν έχει τελειώσει, αλλά είχε μια ολόκληρη διάσταση προς την κατεύθυνση αυτή, χαρτογράφηση και εντοπισμός ευάλωτων ενάλλειων οικοσυστημάτων. Για μένα η δημιουργία ζωνών είναι λύση εν μέρη. Και να επανέλθω με το, στο θέμα αυτό σε κάτι που είχε πει ο κύριος Βίβερ, αν κατάλαβα καλά, αυτά που είπε, ως προς τις εκτιμήσεις των ζωνών στις οποίες έχει, υπάρχει αντίκτυπος, όπως είπα, η μέγιστη, μέγιστη ε, ζώνη για την αλληλεία ήταν 27.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα για τους πυθμένες, ε, για τα, είδη, τα βαθύβια είδη κάτω των 200 μέτρων. 27.000 τετραγωνικά δεν είναι τίποτα, αλλά είναι το 1 εικοστό της επιφάνειας της Βρετανίας. Και μιλάμε για βυθούς κάτω των 200 μέτρων μέχρι 1500 για όλη την, ε, τα 200 μέτρα πηγαίνουν από το Γιβραλτά. τα πέραν των 200 μέτρων γίνονται από, τα, από το Γιβραλτά, Αζόρες, ε, Βρετανία, μέχρι τη θάλασσα του Μπάρεντς φτάνει. Από πλευράς μου υπάρχει, κατά την άποψή μου, υπάρχει αλία βαθέων υδάτων, αλία που δεν χαρακτηρίζεται βαθέων, βαθέων υδάτων και αλία στο βυσκαϊκό κόλπο που ε, δεν είναι βαθύ βιαλία και που παρά τα αυτά είναι, ε, έχει, είναι πολύ παραπάνω από τα 27.000 χιλιόμετρα. Αυτά για την χωροταξική προσέγγιση. Θα δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο. Κυρία Σακάου, για για την ερώτηση της Πορτογαλίδας συναδέλφου. Δεν ξέρω το κόστος του έργου, ξέρω ωστόσο ότι σε ό,τι αφορά τη χρήση των σκαφών μόνο, χρησιμοποιήσαμε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια του έργου, μια άλλη ερώτηση που μου τέθηκε, ξεκίνησε το 2009 μέχρι τώρα η χρηματοδότηση. Τόπα. Ωστόσο, μετά λόγω της κρίσης η χρηματοδότηση για την Ισπανία και για τη Μεγάλη Βρετανία σταμάτησε. Οι Καναδοί που είχαν εμπλακεί και αυτοί συνεχίζουν να χρηματοδοτούν μέχρι το Μάρτιο του 2014 και οι βασικές δομές που χρηματοδότησαν το έργο ήταν η Γενική Γραμματεία για τη Θάλασσα στην Ισπανία, το ΣΕΦΑΣ το Ηνωμένο Βασίλειο και η καναδική κυβέρνηση. Η κατάσταση τώρα έχει ως εξή. Προσπαθούμε, βρίσκεται υπό διαδικασία η έγκριση νέας χρηματοδότησης, αλλά αργή, είναι αργή η διαδικασία. Η Ένωση μέχρι μέσω του ΝΑΦΟ, από ό,τι φαίνεται, θα χρηματοδοτήσει το έργο, ούτω ώστε μέχρι το 2014 τουλάχιστον να ολοκληρωθούν οι αναλύσεις όλων αυτών των ε, διαδικασιών, ούτως ώστε και να προχωρήσουμε και σε εργαστηριακές ε, μελέτες για να δώσουμε τα όρια των πολυγόνων, δηλαδή των κλειστών περιοχών. Για την άλλη ερώτηση, για την ζώνη του ΝΕΑΦ, ο, ο για το έργο αυτό είναι ένα συνάδελφο ο Παόλο Ντουράν που λείπει, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Το έργο αυτό ήταν ε, πρωτοπόρο στο Ισπανικό Οκεανογραφικό Ινστιτούτο. Ήταν το πρώτο έργο που ασχολούσε με τα, που ασχολιόταν με τα ευάλωτα ενάλια οικοσυστήματα το έργο αυτό που έχει παρόμοια μεθοδολογία με αυτή που σας περιέγραψε για το δικό μας τον Ιδίδες, η χαρτογράφηση δηλαδή της ζώνης, πήραμε δείγματα από το βυθό για να δούμε τους οργανισμούς που... Τι, Κλείσαμε 16.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Αλία το 2012. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, μπορώ να μιλήσω με τον Παύλο Ντουράν, που θα σας ενημερώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο, ίσως να μπορέσω να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Κύριε Λοράν, θέλετε να τελειώσετε κάτι. Άλλες ερωτήσεις. Για τον κατάλογο των ειδών. Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε το 12. Δεν ήταν έτοιμα τα κείμενά μας τότε. Υπάρχει, προτείνει η Επιτροπή ένα κατάλογο ειδών με αντικειμενικά κριτήρια όπως σας τα περιέγραψα. Ωστόσο, εμείς ε, προτείναμε διαφορετικό κατάλογο ειδών. Στον τελικό κανονισμό θα υπάρξει φαντάζομαι εν τέλει ένας τελικός κανονισμός ο οποίος θα περιλάβει ενδεχόμενα και θέματα χώρο, ε, διαχείρισης χώρου. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ειδών πάντως, οι προτάσεις μας με, με ποσοτικοποιημένα κριτήρια μπορούν φαντάζομαι να μελετηθούν από την Επιτροπή, είναι έτοιμα τα μελετήσει η Επιτροπή και να βελτιώσει ενδεχόμενα, ενδεχόμενα τις δικές της προτάσεις. Για την ερώτηση του κυρίου Αρσένη, η τελευταία. για το κατά πόσον στο Deep Fishman υπήρχαν τεχνολογίες ε, ε αλλιευτικών ε, εργαλείων. Όχι, δεν είδαμε τα διάφορα εργαλεία. Ευχαριστώ. Προς την Επιτροπή τέθηκαν ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Φρύς, να μας απαντήσει, αν θέλει. Φράγα. Κυρία Φράγα. Άκουσα αυτά που είπε ο εκπρόσωπος του Deep Friesman και βεβαιωμένο ότι δεν υπάρχουν συστάσεις, κάποιες δεν λήφθηκαν υπόψη και η Επιτροπή μπορεί να τις αγνοήσει μήπως θα έπρεπε να περιμένει να τελειώσει το έργο για να κάνει μια τελική πρόταση και να μην χρειάζεται να κόβει ράβη στην πρόταση που άλλα ακούει, άλλα δεν ακούει, παρότι η ίδια ανέφεσε την διεξαγωγή της. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε το πρόγραμμα Deep Fishman είναι ένα από τα διάφορα προγράμματα που βοηθούν πάρα πολύ και όπως ακούσαμε σήμερα κατ' ουσίαν πρόκειται για τη βελτίωση της επιστημονικής βάσης ε, για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων βαθέως ευηθού. Βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε και μία άλλη σειρά ε, συναφών θεμάτων ένα από αυτά τα θέματα είναι η δημιουργία ευκαιριών. Ακούσαμε ε, για νέες μεθόδους εντοπισμού αποθεμάτων. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και όπως γνωρίζετε ε, βοήθησε τα μάλα ε, στον τελευταίο γύρο του Δεκεμβρίου για να λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου σε είπαν, ισχυρίστηκαν πράγματα τα οποία βασίζονται ακριβώ στα ευρήματα αυτού του project. Υπάρχουν και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα. Υπάρχει το θέμα των ε, σημαντικών ειδών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τρία βασικά στοιχεία που προσπαθήσαμε να εξετάσουμε στην πρότασή μας. Πρώτον, το σύστημα αντιοδότησης, το οποίο είναι στοχευμένο στα βαθέα ύδατα. Το δεύτερο είναι ο εξοπλισμός και το τρίτο η συγκέντρωση, η συλλογή δεδομένων. Έτσι λοιπόν αυτά τα τρία θέματα δεν είναι δεν έχουν ε, άμεση σχέση με το πρόγραμμα Deep Fishman είναι αυτόνομα, αλλά υπάρχουν και άλλες μελέτες που λαμβάνουμε υπόψη μας. Ε, έχουμε βρει λοιπόν διάφορα ευρήματα, ορισμένα εξ αυτών, ορισμένα project έχουν ολοκληρωθεί, αλλά συνεχίζονται. Η Κομισιόν κάνει την πορεία για να λάβει υπόψη της ε, τα ευρήματα και με βάση αυτά προχωράμε μερικές φορές πρέπει να δεχτούμε ότι η επιστημονική γνώση προχωράει και κατά τη διάρκεια ε, όσο είμαστε μέσα στη διαδικασία, την νομοθετική. Ε, γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε εδώ για να μάθουμε και αν μάθουμε κάτι ε, συγκεκριμένο για τις προτάσεις μας, είμαστε οι τελευταίοι που θα πούμε ότι πρέπει να αγνοηθεί. Κάθε άλλο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Προχωράμε. Το επόμενο πάνελ. Μελέτης περιπτώσεων Γαλλία-Πορτογαλία. Η κυρία Κλέρ Λουβιάν. Thank you very much. Um, so I'm going to just uh, go through a brief historical overview. Μια ιστορική μελέτη. Ε, κοιτάξτε να δούμε λιγάκι αυτά τα θέματα ε, των βαθιών και κατόπιν τη εντράσεις αγοράς. Το Bloom είναι μη κερδοσκοπικό οργανισμός. Έχουμε δημοσιεύσει το βιβλίο μας σε 11 γλώσσες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης ε, οργανώσαμε και μια έκθεση που πήγε σε αρκετές χώρες. Ε, μέχρι τώρα είχε χίλιους ε, επισκέπτες στο Χονγκ Κόνγκ, στο Παρίσι. Εκεί βρισκόμαστε και είμαστε μέρος του συνασπισμού που αποτελείται από 70 ΜΚΟ και έχουν ως στόχο την προστασία του ωκεανού από καταστρεπτικές δραστηριότητες. Μας ενδιαφέρει να έχουμε βιώσιμες πρακτικές, να διαφυλάξουμε διάφορα είδη ε, και να υπάρχει και ένα είδος ε, διαχείρισης ε, δημόσιων κονδυλίων. Επίσης, μας ενδιαφέρει το θέμα της παιδείας. Συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις όπως με την Κινέζικη, τη Γαλλική και διεξάγουμε και ανεξάρτητες έρευνες. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη που δείχνει τη σημασία που έχει κάθε χώρα. Ε, πρόκειται για τη σώρευση ειδών βαθέων υδάτων μέσα από τα χρόνια. Αυτό ξεκίνησε δεκαετία του 60 και του 70 για τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλού όμως ξεκίνησε νωρίτερα. Η Γαλλία βρίσκεται στην 7η θέση μετά τη Νέα Ισλανδία, την Ισλανδία, τη Ρωσία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Η ε, αλία σε βαθέιδατα των Γάλλων ε, εδώ ε, αναφέρομαι και σε αυτά που είπε ο κύριος Λορόν, τα είπε πάρα πολύ καλά. Η έναρξη αυτής της ελίας ε, ξεκίνησε ως ε, αποτέλεσμα της υπερελήψης αποθεμάτων στη Βόρεια Θάλασσα και στον Βόρειο Ανατολικό Ωκεανό. Δυστυχώς προέκυψε μείωση των παραδοσιακών αποθεμάτων όπως είναι το βατραχόψερο και η πεσκανδρίτσα. Έτσι λοιπόν ε, υπήρξε μία ανακατανομή της αλίας, ε, απλωθήκαμε και σε βαθέα ύδατα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο για την εκμετάλλευση της ε, θάλασσας, το Ινστιτούτο αυτό ε, προσπάθησε να βρει νέους ε, χώρους για την Αλία, στο Ρόκελν Χάτν και σε άλλες περιοχές, ε, στον Βόρειο Ανατολικό Ωκεανό. Έτσι λοιπόν οι ε, προσπάθησαν απεγνωσμένα να βρουν νέα αλληλευτικά αποθέματα. Στη Γαλλία υπήρξε μία αγορά Βέβαια τα ψάρια αυτά που ε, ψαρεύαμε δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικά, γι' αυτό άλλαξε, άλλαξε η ονομασία τους. Ε, ε Παραδείγματος ε, χάρη το σλάμινγκ το μετανομάσαμε, το είπαμε ψαρό του Ατλαντικού Orange Ruffy στα αγγλικά. Τέσπα ονομασίες που να είναι πιο αποδεκτές από τους καταναλωτές. Οι Αλείς επίσης ε, είπαν στους ε, κατανοητές ότι πολλά αυτά τα ψάρια θα τους τα έδιναν δωρεάν αν δεχόντουσαν τα νέα τους ονόματα. Η μεγαλύτερη κατανάλωση που υπάρχει στη Γαλλία και στις ε, δυτικές περιοχές αφορά αυτά τα ψάρια. Βλέπετε σε αυτό το γράφημα ότι τα περισσότερα ψάρια όπως ο μαύρος μπακαλιάρος και το βατραχόψαρο, αυτά ε, προήλθαν από ε, βαθέα ύδατα και όπως σας είπα προέκυψαν επειδή υπήρξε ε, μείωση των παραδοσιακών αποθεμάτων. Στη Γαλλία έχουμε μια ειδική κατάσταση. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία ε, του 10 και βλέπετε ότι το 83% των αλλιευμάτων βαθέων υδάτων ε, της ε, Γαλλίας βλέπουμε ότι το 83% αποτελείται από τρία βασικά είδη. Αυτό είναι το 83%. Κατόπιν το καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού. Υπήρξε μια επιδρομή αυτού του ψαριού και σε προηγούμενο γράφημα είδαμε ότι δυστυχώς μειώθηκε κατά πολύ το απόθεμά του. Έτσι λοιπόν ε, τα ψάρια αυτά ε, δεν ήταν ελκυστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από το 1998 βλέπουμε μία αναδιοργάνωση των στόλων για να διασφαλιστεί ότι ό,τι αλίευαν στον Βορειοατλαντικό ωκεανό θα έφταναν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία για να αποφύγουν το κόστος του να πάνε στη Γαλλία. Ήταν πολύ ακριβά τα καύσιμα και ο χρόνος βέβαια. Οι Γάλλοι, οι γαλλικοί στόλοι Υπάρχουν στοιχεία από το Υπουργείο Γεωργίας και από εθνικούς ε, φορείς ε, που προάγουν την αλία στη Γαλλία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 89 41 σκάφη ασχολούνται με την αλία βαθέων σκαφών και μόνο 6 εξειδικευμένα σκάφη. Μέχρι το 85. Μετά 58 σκάφη για βαθέα ύδατα και 20 πλέον εξειδικευμένα σκάφη και αργότερα το 2010 βλέπουμε ότι έχουμε μέχρι 30 ειδικέ άδειε και 11 εξειδικευμένε μονάδες. Το 90 περίπου αυτών των μονάδων από αυτά ε, προκύπτει ότι κάτω από 10 τόνους είναι τα ψάρια από τα βαθιά Άρα δηλαδή οι Γαλλίες έχουν κάποιες, οι Γάλλοι έχουν κάποιες ε, ειδικέ άδειε ε, που τους επιτρέπουν να λεύουν στα βαθιά αλλά είναι περιορισμένες οι ποσότητες. κατεβλήθησαν προσπάθειες ε, για να κατηγοριοποιηθούν τα σκάφη. 11%, 11 σκάφη ε, ψαρεύουν τις μεγαλύτερες ποσότητες. Ε, βλέπετε λοιπόν εκεί στη διαφάνεια που δυστυχώς εμείς οι διερμηνείς λυπάμαι αλλά δεν βλέπουμε. Βλέπετε λοιπόν τα σκάφη ε, τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την αλία βαθεών υδάτων. Οι αλλαγές είναι οι εξής. Το 2000 είχαμε μια λυσίδα που έχασε ένα σκάφος με ένα ατύχημα στην Ιρλανδία. Ένας άλλος στόχος, στόλος, γαλλικός πάντα, σκάφη γαλλικά, μετατράπηκαν σε εξειδικευμένα σκάφη πλήρους απασχόλησης, ε, πλέον ε, αυτός ο στόλος ε, αλλιεύει τον ε, μαύρο μπακαλιάρο και πολλάκα και πολλά λοιπόν από αυτά τα σκάφη όπως σας είπα ασχολούνται πλέον με την αλία σε βαθαία σκάφη, σε βαθαία ύδατα. Τρία όμως είναι πλέον τα οποία αλεύουν περισσότερους από 500 ε, τόνους το χρόνο. Τα ε, είδη βαθέων υδάτων πλέον ε, αντικατοπτρίζουν ή αντιστοιχούν στο 40 περίπου του ε, συνολικού όγκου των μεγάλων τρατών. Ίσως να έχει αυξηθεί η ποσότητα γιατί υπάρχουν πλέον υπάρχουν ανακατανομές ε, των ποσοτήτων και αυτές οι δύο μεγάλες ε, τράτες ε, μοιράζονται μεταξύ τους την ποσότητα. Πρέπει λοιπόν ε, να πούμε ότι το 40% των ε, αλλιευμάτων αυτών των ε, σκαφών αφορούν, το 40% αφορά είδη βαθέων υδάτων. Οι εταιρείε και αυτή συγκεκριμένη στην οποία αναφέρομαι, κατά 60% αλλιεύει σε βαθέα ύδατα αλλά το ποσοστό μπορεί να αναβαίνει και σε 86%. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτη στην αγορά. Τα supermarket Intermarché γιατί ασχολούνται αυτά με την αλία. Βέβαια αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτή η αλυσίδα σούπερ έχει μια κάθετη πολιτική ε, και γι' αυτό λοιπόν τον λόγο ο πρώην διευθύνων σύμβολος ε, είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση ε, στις πρώτες ύλες στον αρχικό εφοδιασμό. Υποτίθεται ότι θα υπήρχαν έρευνες για να διαπιστωθεί κατά πόσον η αλληλεία με την, την οποία αναπτύσσουν είναι οικολογικά συμβατή. Υπήρξαν βέβαια αρκετά προβλήματα. Κατόπιν τούτου η μελέτη ε, που δημοσιεύτηκε ήταν ε, πολύ δυσάρεστη για την κυβέρνηση ε, γιατί δεν υπάρχει καμία αναφορά και η μελέτη που έγινε με παρεμφερεί άλλες μελέτες δεν έχει συμπεριληφθεί. Κατόπιν τούτο ο φάκελος αυτός ε, δεν έχει νομική τεκμηρίωση. Πάντως ε, όλα αυτά υπάρχουν ε, στο διαδίκτυο, στα αγγλικά αν θέλετε να τα μελετήσετε. Η διαδικασία όμως κατέδειξε ότι αυτοί όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί παράμετροι παρακάμφθηκαν και θεωρήσαμε ότι άξιζε τον κόπο να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε και να συγκεντρώσουμε στοιχεία. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Έχουμε αυτή τη διαφάνεια ε, σχετικά ε, με την προσέγγιση και τις εκτιμήσεις για τις θέσεις εργασίας. Ε, δύσκολο είναι βέβαια αυτό αν δεν έχει κανείς αδειάσει στα στοιχεία. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτή την ε, συγκεκριμένη μας αποστολή μιλάμε για 100 μέχρι 200 θέσεις απασχόλησης και η Κομισιόν όταν δημοσίευσε τη δική της την έκθεση σχετικά με τις ε, τράτες μιλάει για 600 ε, θέσεις σε σχέση με τη Γαλλία. Διερωτώμεθα λοιπόν πώς γίνονται οι υπολογισμοί Κάναμε σχετικές ερωτήσεις, αλλά δεν μας δόθηκαν οι απαντήσεις. Και κατόπιν του ε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε ε, ουσιαστικά. Στην εταιρεία Σκαρπές ε, γίνεται λόγος μόνο για εννέα σκάφη. Τα έξι όμως ε, είναι για βαθαία ύδατα. Κάτι άλλο που κάναμε είναι ότι βασίσαμε την ανάλυση μας σε λογαριασμούς, γιατί εκεί ε, δεν μπορεί κανείς να μπερδέψει τα στοιχεία. Το μόνο μπορεί να κάνει να ε, σχολιάσει τα στοιχεία. Το 2011 δημοσιεύσαμε μία ανάλυση και θελήσαμε να ενημερώσουμε τα βασικά ευρήματα που ήταν τα εξής. Οι τρεις ε, μεγαλύτεροι στόλοι που ασχολούνται με αλία βαθέων υδάτων έχουν επιδοτηθεί η ε, Σκαρπές δεν δημοσιεύει πλέον τους λογαριασμούς της από το 2009 και γι' αυτό το λόγο ε, καταφύγαμε σε νομικές συμβουλές. Τους πείσαμε ε, να δημοσιεύουν πλέον τους λογαριασμούς τους και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούν αυτούς τους λογαριασμούς, τους οποίους όπως σας είπα αποκτήσαμε μετά από την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων. Από το 2006 μέχρι το 2011 ε, έλαβαν ε, επιδοτήσεις 4,9 εκατομμυρίων ευρώ και από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη Γαλλία. Το ίδιο ισχύει και για την Σκαρπές με βάση τους λογαριασμούς που έχουν δημοσιεύσει. 9,5 περίπου τα εκατομμύρια ευρώ που έλαβαν και η DLM έλαβε ε, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ ε, με τη μορφή επιδοτήσεων. Μπορούμε λοιπόν να δούμε λιγάκι τα οικονομικά αποτελέσματα. Έχω να. Έχει σωρεύσει 8,1 εκατομμύρια ευρώ ε, καθαρή ζημιά παρά την ε, επιδότηση. Αυτοί λοιπόν κατ' ουσίαν ε, καταστράφηκαν και βλέπουμε ότι από τότε που τους εξαγόρισαν οι UK Fisheries ε, και κατ' ουσίαν αποδεσμεύθηκαν από την αλία σε βαθιά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση στην κατάστασή τους. Σκαρπές τώρα. Ε, σημειώνουν και αυτή η ζημιά στο ίδιο χρονικό διάστημα, αποφορολογημένη ζημιά, παρά τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, παρουσιάζουν ε, και αποπληρωμές δανείων τα οποία είχαν λάβει. Άρα δηλαδή η πραγματική ζημιά, αν δεν υπήρχε η δανειοληψία, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Η έχει και αυτή η καθαρή ζημιά, εμφανίζει η καθαρή ζημιά ε, και αυτά ε, αποφορολογημένα και 7 εκατομμύρια ευρώ είναι το οικονομικό αποτέλεσμα ε, και ένα απρόβλεπτο κέρδος. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται στη διαφάνεια και φαίνεται εκεί ότι υπάρχουν κινήσεις για να βελτιωθεί η δική τους η κατάσταση. Τώρα, δείκτης απόδοσης και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια που θέλω να προβάλλω. Πραγματικός δείκτης απόδοσης ε, είναι ε, τα λειτουργικά αποτελέσματα. Τζίρος μείον παγίων δαπανών, μείον πάγιες δαπάνες. η ογνώ βελτιώθηκε και τώρα πλέον παρουσιάζει κέρδος. Άρα δηλαδή η αλληλευτική δραστηριότητα είναι επικερδής. Δεν είναι μεγάλο το κέρδος, είναι του 2% αλλά τουλάχιστον δεν παρουσιάζει έλλειμμα. Οι σκαρπές ε, και αυτή βρίσκεται περίπου στην ίδια κατάσταση. Αν δούμε την Delum, το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι 25%. Αυτό είναι ένα ποσοστό του κύκλου εργασιών. Όταν λέμε λοιπόν ότι μια ληφτική εταιρεία χάνει το 25% με τη μορφή λειτουργικού αποτελέσματος, αυτό σημαίνει 25% στο τζίρο. Άρα δηλαδή η αλληλευτική δραστηριότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι μόνο επικερδής, αλλά δεν είναι καν βιώσιμη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ντελέμ, αν δεν έχει ήδη ε, καταρρεύσει, σύντομα ε, θα τεθεί προς πώληση. Και έχω άλλη μία διαφάνεια για την αντίδραση αγορά στη Γαλλία για να σας δείξω ότι ορισμένα σούπερ μάρκετ ε, πλέον ε, ε, δεν πουλάνε ψάρια βαθέων υδάτων. Αλλά κατ' ουσίαν αυτά είχα να σας πω στην ομιλία. Ναι, ναι, ναι. ευχαριστώ. Λυπάμαι, αλλά έχουμε περιορισμένο χρόνο. Ο λόγος στον κύριο Λιμπεράτο Φερνάντες. Ε, Γεια σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας αποφθήνατε. Ευχαριστώ, λέω, για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. για τις ε, απαιτήσει σε πρόσβαση σε είδη βαθέων ε, υδάτων. Αντιπροσωπεύω ε, την, τον Επαγγελματικό Σωματείο των Αλλιέων του Πόρτου Ντεαβρίγου στις Αζόρες. Είμαστε οργάνωση παραγωγών, αναγνωριστήκαμε το 1993, παρόλο που είχαμε δημιουργηθεί το 1976, πριν την είσοδο τη Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε με ένα στόλο με μικρέ διαστάσει, μόνο τέσσερις από, τέσσερα από τα μέλη μας έχουν ε, σκάφη των 30 περίπου μέτρων ε, με ικανότητα να ψαρεύουν στα ανοιχτά ύδατα. Πάνω από το 80% ε, των σκαφών μας είναι πολύ μικρά, ε, δύο μέτρων και προφανώς δεν μπορούν να περάσουν να σε, στα ανοιχτά πέρα των δύο μιλίων. Πάνω από το 70% των αλλιευμάτων ε, είναι ε, βαθύβια ε, ψάρια. Βρισκόμαστε σε κρίση και η αλία δίνει ψωμί περίπου στο 60% του ενεργού πληθυσμού στις Αζόρες. Από αυτούς το 40% είναι εγγεγραμμένοι αλείς, αναγνωρισμένοι αλείς και ε, το 60% ε, του συνολικού τομέα ε, είναι συναφείς δραστηριότητες, είτε πρώτης αλίας για την προετοιμασία της αλίας, είτε στη μεταποίηση κλπ. Στη, στα κονσερβοποιεία, τα οποία δεν ασχολούνται με βαθύβια ψάρια, δουλεύουν κυρίως με γυναίκες. Θα περάσω τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Ήθελα να σας δείξω μια εικόνα που να αντιπροσωπεύει την αλία ε, όλου του Ατλαντικού μέχρι τη Μικρονησία. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Ε, το, μεταξύ 2004 2007 συμμετείχαμε στην δημιουργία του ΡΑΚ και στην ομάδα εργασία ε, παρακολούθηση τη Αλία στα νησιά. Αυτό μα επιτρέπει να ε, δούμε τι διαφορέ που υπάρχουν ανάμεσα στη Μαδέρα, τα Κανάρια και στι ε, Αζόρε. Και οι τρει βέβαια, τρει περιοχέ είναι στο, μέσα στον Ατλαντικό και δεν έχουν φαλοκρηπίδα. Ε, τα βασικά μας ε, είδη όπως το σπαθόψαρο και το τόνος ε, έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Παρόλο ότι τα ύδατά μας είναι πολύ, μια πλωτή, πολύ πλατιά περιοχή, αντιπροσωπεύουν το 80% της ΑΟΣ της Πορτογαλίας, το, τα αλλιεύματά μα αντιπροσωπεύουν μόνο το 6-8% τη ε, ε, παραγωγής, ε, της εθνικής παραγωγής στις ενώ στη Μαδέρα το 2-3% τη εθνική παραγωγή. Αυτό αποδεικνύει ε, την, το ευαίσθητο της περιοχής ε, ε, σε βιολογικό επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία αλλά μια πολύ μικρή παραγωγικότητα, 10% περίπου οι ενευτικές περιοχές ε, βρίσκονται, είναι παράκτιες ε, στα τρία μίλια από την ακτή και ε, ενώ έχουμε πολλές ευαίσθητες περιοχές έξω από αυτή τη ζώνη. Η αλληλεία σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα στις Αζόρες, μπορούμε να πούμε ότι έχει μια διπλή εξάρτηση εξαρτάται αφενός από τη, τα βαθύβια είδη και από τη, το γεγονός ότι είναι σχεδόν μοναδική η δραστηριότητα για τα νησιά, τουλάχιστον μία από τις πολύ λίγες οικονομικές δραστηριότητες. Έχουμε ένα πίνακα μέσω του οποίου μπορείτε να διαπιστώσετε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε μείωση των αλληλευμάτων ε, ε, και μείωση της, ε, του εισοδήματος, της αξίας τους. Ε, η ο στόλος μας ε, για τον τόνο ε, αποτελείται από 20 σκάφη ε, και αλλιεύουν και στη Μαδέρα και στις Αζόρες. Έχουμε πάνω από 100 βαθύδια ζώα, είδη, αλλά οι ταλεύματά προέρχονται από πολύ ε, λίγα ε, ε, είδη. Ε, μπεριτσίδες, ε, το σπαθόψαρο, το, το σπαθόψαρο ειδικά ε, είναι σε, σε πειραματική φάση. Στις Αζόρες, ενώ στην Μαδέρα αντιπροσωπεύει το 55% στο 60% των λιευμάτων που πολλούνται. Δηλαδή στην Μαδέρα ε, η, τα βαθύ διαλύα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από αυτό το είδος. Ε, το, η αλία λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες ε, ε, επηρεάζει τα, τα οικοσυστήματα, επηρεάζει αρνητικά πολλά θαλάσσια οικοσυστήματα όπως τα κοράλια και όταν οι αλληλείς ε, ψαρεύουν με τράτες βυθού, ε, ε φτάνουν μέχρι το βάθη των 2.000 μέτρων. Ε, δεν υπάρχουν ποσοστώσεις σε αυτά τα ύδατα και ότι ε, ό,τι αλλιεύεται μπορεί να πουληθεί. 60 περίπου είναι τα σκάφη στις Αζόρες. Ε, όμως, 220 ε, τόνοι παραγωγής χάθηκαν ε, εξαιτία ε, του κλεισίματος μιας περιοχής που είναι σε διεθνή ύδατα και αυτό αποτελεί σημαντικό πλήγμα. Ε, ταυτόχρονα υπάρχουν ρωσικά πλοία και από τις ε, πλοία από τις νήσες Φαρόες που ε, αλλιεύουν ε, χωρίς κανόνες. Ε, και ορισμένα σκυλόψερα βυθού και ορισμένα σπαθόψερα ε, και άλλα είδη, οτιδήποτε αλλιεύεται σε διεθνή ύδατα, ε, αλλιεύεται από σκάφη άλλων χωρών χωρίς ε, κανόνες. Η, η πυρωτική αλία στην Πορτογαλία εξαρτάται σε ένα βαθμό από τα ε, μαθήβια είδη. δεν έχουμε όμως στράτες βυθού κατά βάση. Αλλά στην Ζεζίμπρα που είναι ένα από τα σημαντικά λιμάνια της Πορτογαλίας, εξαρτάται όλο το λιμάνι από, την, από το σπαθόψαρο. Θα ήταν σημαντικό να διαθέτουμε κανόνες για όλο τον Ατλαντικό και το Βόρειο Ατλαντικό από τα Κανάρια μέχρι το Βορρά. Ε, αυτοί οι κανόνες ε, θα πρέπει να αφορούν και είδη τα οποία είναι παρεπίπτοντα. Όπως για παράδειγμα ορισμένα είδη ε, ψυχιλόψαρου. Τα στοιχεία που διαθέτουμε αποδεικνύουν ότι η αναπαραγωγή γίνεται στα νότια της ζωρών, για παράδειγμα για το σπαθόψαρο μεταξύ Μαδέρας και Αζωρών, η, τα σκυλόψαρα από την άλλη μεριά ε, σε, στα ύδατα του βόρειο-ανατολικού Ατλαντικού. Οπότε εμείς υποστηρίζουμε τη συμπερίληψη στον κανονισμό συγκεκριμένων απαιτήσεων για τα βαθιά ύδατα για όλο τον βορειοανατολικό Ατλαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και το Συμβούλιο, θα πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα που θα εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη, αλλά και ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να πιστούν και τα Ηνωμένα Έθνη να ε, επιβάλλουν κανόνες για τα πλοία άλλων χωρών, τρίτων χωρών που αλλιεύουν στα ίδια ύδατα. Σε ό,τι αφορά τι στράτε βυθού, οι Αζόρες έκαναν ένα πείραμα το 2001-2002 για, ε, με, ένα, με μια τράτα νεοζιλανδέζικη. Ε, ε, βάλαμε δύο δικού μας ναυτικούς πάνω σε αυτό το πλοίο και διαπιστώσαμε ότι οι πρακτικές που εφάρμοζε ε, ήταν ε, πολύ κακές και για το βυθό και, για τα και λόγω παρεμπιπτών των αλλιευμάτων. Μετά από αυτό το πείραμα, μετά από αυτή την εμπειρία, ε, ε, ψάρμαν κυρίως ε, καθρεπτό ψαρό, ε, εμείς μετά από αυτήν την εμπειρία είδαμε ότι 7 ε, τόνοι ε, σπαθόψαρου είχαν αλλιευθεί ε, ως παρεπίπτον αλλιεύμα. Οπότε όσο προσεκτικά και να γίνει, η αλλίευση μετρά τα βυθού έχει αρνητικές επιπτώσεις. Δεν είναι βέβαια δυνατόν να καταρριχθεί μια δραστηριότητα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στη βιωσιμότητα, να έχουμε ένα πρόγραμμα μείωση τη αληθική προσπάθεια. Και για τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα σκάφη τρίτων χωρών. Θα πρέπει η ΦΑΟ, η ΚΟΦΗ, ε, οι, οργανισμοί, οι φορεί των ΗΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν παρόμοιο πρόγραμμα για να καταργηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον ε, αυτού τύπου η αλία γιατί οι επιπτώσεις ε, επί των αποθεμάτων, των αποθεμάτων είναι πιο αρνητικές από θετικές. Για παράδειγμα, 600 σκάφη, 3.000 αλίες. Ε, έχουμε αλία μικρής ε, κλίμακος. ενώ κάποιοι οι οποίοι ψαρίνουν στα βαθιά υδατά δεν έχουν καμία σχέση με, την, με τη γη με το νησί, με τη στεριά. Ε, αυτοί πηγαίνουν εδώ σήμερα και, και αλλού αύριο. Εμείς ψαρεύουμε πάντοτε δίπλα στα νησιά μας και γι' αυτό το λόγο ε, είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί με τα οικοσυστήματά μας. Λοιπόν, ε, το, το επάγγελμά μας ε, ε, μας εξασφαλίζει πολύ χαμηλό εισόδημα έχουμε πληγεί πάρα πολύ από τη μείωση των ε, αλλιευμάτων. Και παρόλο ότι εμείς υποκείθεμεθα σε ελέγχους και κανόνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντέκ έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους δύο παρεμβαίνοντε, την κυρία Νουβιάν και τον κύριο Φερνάντε, για τι παρουσιάσει του. Ωστόσο, δεν θα σας εκπλήξει, θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Στην κυρία Νουβιόν κυρίως. Δεν φαντάζομαι την εκπλήσει. Κυρία μου, δεν, είναι, δεν ήθιστε εδώ να κατηγορούμε συγκεκριμένα και ονομαστικά επιχειρήσεις. Όπως διαπιστώσατε από το ξεκίνημα της ακρόασης, οι ειδικοί μα ε, κάνουν γενικέ παρατηρήσει, αν μη τι άλλο. Δεν σα διέφυγε, νομίζω ότι εδώ δεν είναι ούτε εισαγγελία, ούτε δικαστήριο. Έτσι όπως σας άκουγα, είχα την εντύπωση ότι ερχόσασταν και δίνετε μαθήματα. Βεβαίω, ανέμενα από πλευρά σα ε, ένα κατηγορητήριο κατά τη γαλλική αυτή εταιρεία, που δεν θα αναφέρω εγώ. Δεν εκπλήσει λοιπόν Ειλικρινώς ωστόσο πίστευα ότι θα μας δίνατε και άλλα επιχειρήματα. Έρχεστε και κάνετε μια λογιστική ανάλυση και πρέπει να είστε πολύ καλή λογίστρια, αλλά τέλος πάντων στη λογιστική ανάλυση έχετε κάποια μεροληψία ή τέλος πάντων είναι αμφισβητούμενοι. Ε, ευρέως θα έλεγα. Και τελειώνοντας, να σας πω ότι δεν πιστεύω, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η εταιρεία αυτή μόνο φιλανθρώπους περιλαμβάνει. Δηλαδή, βγάζουν πλοία για να χάνουν. Μόνο για να χάνουν. Και ε, για το σκοπό αυτό απασχολούν εκατοντάδες προσωπικό. Αν αυτό συμβαίνει πραγματικά κάτι δεν καταλαβαίνω. Σας το είπα και σε προσωπική συνάντηση που είχαμε. Μιλάμε για επιχειρηματίες που προφανώς θέλουν να βγάλουν κέρδη. Η, από ό,τι γνωρίζω η εταιρεία αυτή έχει κέρδη. Η ανάλυση σας λοιπόν αμφισβητείται ευρέως. Αυτό είναι το λιγότερο μπορώ να πω. Μπορεί να μιλάμε όλο το βράδυ αν θέλετε, αλλά θεωρώ κρίμα που στο χώρο αυτό επιτίθεστε σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Σύντομα να είστε, γιατί δυστυχώς ο χρόνος δεν πάει καλά, εξαιτία μου. Κύριε Τωμά, ευχαριστώ. Λυπάμαι από αυτά που άκουσα από την κυρία Νούβιον. Όχι, δεν με εκπλήσει, διότι προφανώς ήρθε εδώ πέρα για να καθαρίσει τους λογαριασμούς της με μια γαλλική επιχείρηση που είναι και από την περιοχή μου. Ωστόσο, και πραγματικά δεν ξέρω πώς οργανώσαμε την ακόραση αυτή. Αν θέλαμε να υπάρχει μια κοινωνικο-οικονομική ανάλυση και μια παρατήρηση για τις καπιταλιστικές ε, αποδόσεις των επιχειρήσεων, καλύτερα θα ήταν να το κάνει οικονομολόγος. Πόσο μάλλον που η ακρόαση που παρουσίασε είναι γεμάτη σφάλματα. Εγώ, ούτε οικονομολόγος είμαι, ούτε ξέρω τις επιχειρήσεις αυτές, ξέρω καλύτερα τα στοιχεία. Δύο παραδείγματα σας δώσω. Πρώτον, οι ενισχύσεις για, τις, ε, για τις, ε, τα δηληστήρια αυτά ε, ήταν ενισχύσεις που έδωσε η Γαλλία σε όλες τις... η ενισχύσεις για το δίζελ, συγγνώμη, ε, ήταν ενισχύσεις που έδωσαν σε όλες τις επιχειρήσεις Γαλλίας στα πλαίσια της κρίσης του 2009. Άρα δεν αφορούσε συγκεκριμένα σκάφη. Λοιπόν, ήρθε για να καθαρίσει τους λογαριασμούς της και μας λέει και λάθη. Είναι δυνατόν να γίνει μία μελέτη για τον αντίκτυπο του σχεδίου κανονισμού για να ξέρουμε τουλάχιστον πόσα είναι τα εμπλεκόμενα σκάφη και τι, ποιος είναι ο κοινωνικονομικός αντίκτυπος του έργου αυτού. Θα σας υποστηρίξω, λέει ο κύριος Άγνιο, παρότι είμαι Βρετανός, γιατί δίνουμε του κόσμου τα λεφτά στην Ένωση, όπως ξέρετε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που είπατε ήταν πολύ ενδιαφέρονα. Ανοίξατε το καπάκι, μην το ξανακλείσουμε. Υπάρχουν στη Γαλλία ε, βουλευτές που θέλουν να επανέλθουν ενισχύσεις, ε, ε, κρατικές ενισχύσεις σε ανθρώπους για να πάνε να λαιλατίσουν τους ωκεανούς. Τι, τι, τι είναι αυτό. Μια εταιρεία ζητά ενισχύσεις και θέλει κέρδη. Πώς, έχετε υπολογίσει πόση είναι η ενίσχυση ανά άτομο που εργάζεται εκεί. Άλλη ερώτηση. Έδειξε μια στρεβλή εικόνα του κόσμου με τις χώρες, μια, μια στρεβλωμένη εικόνα του κόσμου με τις χώρες μεγαλύτερες, τις χώρες που έχουν μεγαλύτερη αλίευση. Αυτό τι είναι, ανά άτομο, ανα, ανα ή είναι το σύνολο της χώρας. Γιατί βλέποντας τις Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι όπως φαίνεται είναι, δεν έχει καθόλου αλληλευτική βιομηχανία, αλλά έχει. έχει. Πώς, πώς το λάβατε υπόψη αυτό. Ο Αλά και η Ιζαμπέλ δεν άκουσαν τα ίδια πράγματα και, εγώ δεν ακούσαμε τα ίδια πράγματα και προφανώς δεν καταλάβουμε τα ίδια πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε αφενός έναν οικονομικό κλάδο, την αλία, στη βαθύβια αλία που στο, στη Γαλλία είναι το παράδειγμα, αλλά και σε άλλες χώρες μπορούμε να βρούμε τα αντίστοιχα παραδείγματα που είναι στην εμπροσοφυλακή εκεί, έναν στενό τομέα. Κάποια σκάφη, κάποιες δεκάδες επιχειρήσεις και μία αμφιλεγόμενη τουλάχιστον οικονομική δραστηριότητα που στηρίζεται σε επιδοτήσεις. Τώρα αν είναι επιδότηση δίζελ ή οτιδήποτε το βλέπουμε. Τα στοιχεία που είναι στοιχεία των επιχειρήσεων. Μπορεί οι επιχειρήσεις αυτές να κάνουν κέρδη αλλά δεν αποτελούν κινητήρες της οικονομίας. Είναι ένας κλάδος περιορισμένος με λίγους ψαράδες, μικρή οικονομική δραστηριότητα και από την άλλη ο ίδιος κλάδος παρουσιάζει σοβαρότατες απειλές για το ενάλιο περιβάλλον και τα βαθύβια ήδη ακόμα και τα εμπορικά ήδη που μας αναφέρθηκε προηγουμένως ότι απλά καταφέραμε να σταματήσουμε την μείωσή τους. Με εντυπωσιάζει η δυσαναλογία των ε, θεμάτων. Αυτό πρέπει να το, έχουμε, να το καταλάβουμε. Πέραν αυτού νομίζω ότι η επιλογή μας δεν έχει καμία αντιφατικότητα. Η κυρία Φράγκα. Δεν θα παρενέβαινα, αλλά τώρα μετά από άκουσα πρέπει να παρέμβω. Πρώτον, Πράγματι, και η κυρία Τόμας έχει δίκιο. Ένα από τα προβλήματα που έχει η αξιολόγηση αντικτύπου ε, αυτής της πρότασης Κομισιόν είναι ότι είναι ποιοτική αλλά όχι ποσοτική. Οπότε δεν έχουμε κανένα είδου ε, συγκεκριμένο στοιχείο ποιου στόλου επηρεάζει, ποιε είναι, είναι, είναι οι οικονομικέ επιπτώσει κλπ. κλπ. Οπότε πράγματι να γίνουν γνωστέ οι επιδοτήσει κλπ. Αλλά να προσδιοριστεί να προσδιοριστούν όλες οι επιπτώσεις αυτής της ε, πρότασης, όχι μόνο οι επιδοτήσεις και η Κομισιόν δεν το έκανε. Δεύτερον, σε όσα είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, δεν είναι δυνατόν να μιλούμε μόνο για τις ε, επιπτώσεις στον ελευτικό στόλο, γιατί η πρόταση αυτή έχει επιπτώσεις ε, και σε ό,τι αφορά τα παρεμπίπτοντα λιεύματα, γιατί εκεί ε, επηρεάζεται πολύ μεγαλύτερο στόλο. Ε, συνεπώς, ας μην περιοριζόμαστε. Ε, μην προσδιορίζουμε την, ε, την, ε, τις επιπτώσεις μόνο στα συγκεκριμένα αλλιεύματα. Διότι έχουμε ε, στόλους, πολύ μεγαλύτερους στόλους που επηρεάζονται εξαιτίας των παρεμπιπτών των αλλιευμάτων. Ε, ας γίνει μια κοινωνικο-οικονομική επίπτωση όλων των ε, τομέων που θα επηρεαστούν. Και εκεί να μπουν όλα όσα θέλετε να μπουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεπώ, κύριε Μπεσέτ, ε, το θέμα είναι πολύ πιο πλατή από αυτό το οποίο αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Ε, Κοιτάξτε, θέλω να δώσω μόνο μία πολύ σύντομη απάντηση στην κυρία Φράγκα διότι ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία στη μελέτη αντικτύπου. Και εγώ παραθέτω από τη μελέτη η Γαλλία δύο εταιρείε που ασχολούνται με τη βαθύ διαλύεια, 300 αλληλείς ε, και τα σκάφη τους ασχολούνται με την αλία αυτή. Όσον αφορά την Ισπανία, η Ισπανία δεν έχει καταθέσει στοιχεία, παρότι βέβαια τη τα ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Señor porque es la κύριε Λουβιά. Κοιτάξτε, βλέπω από τις αντιδράσεις ότι ε, προφανώς ε, εμείς ε, αναφέραμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γιατί αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις. Θέλω λοιπόν να πω στα γαλλικά, αν μου επιτρέπετε. Ε, στον κύριο Καντέκ, καταλαβαίνω ότι δεν είναι επιθυμητό να αναφέρουμε συγκεκριμένα ονόματα. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο θα το κάναμε. Αλλά είναι σχεδόν μονοπόλιο. Είναι ε, δεσπόζουσα η θέση του, της συγκεκριμένη εταιρεία. Και φαίνεται ότι αυτή η εταιρεία ε, είναι 100% διοκτησία ενός σούπερ μάρκετ. Και επειδή ε, εμπλέκονται πολύ σημαντικά ποσά με τη μορφή επιδοτήσεων, καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνούμε. Ίσως δεν είναι ότι πρώτη τελευταία φορά αλλά ε, μου φαίνεται ότι αν θέλουμε να ε, έχουμε συγκεκριμένα βάσιμα στοιχεία, διαφανή στοιχεία, θα πρέπει να αναφερθούμε ε, σε συγκεκριμένα ονόματα. Πρόκειται για τους δικούς μας φόρους, όχι μόνο τους γαλλικούς, τους ευρωπαϊκούς φόρους, οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα. Ίσως δεν καταλάβατε γιατί από τη μια ε, μεριά έχουν ζημιές, από την άλλη μεριά ε, η επιχείρηση δεν έχει κλείσει. Να σας πω πολύ καθαρά. Ε, το κέρδος θα πρέπει να επιτυχάνεται σε επίπεδο ομίλου και όχι σε επίπεδο στόλου. Είναι δυνατόν μία επιχείρηση ενός ομίλου να είναι ελληματική, αλλά να επιτρέπει στον όμιλο ή σε μια άλλη επιχείρηση του ομίλου να κάνει πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Μπορεί επίσης για λογιστικούς λόγους ή για φορολογικούς λόγους να επιθυμεί τη διατήρησή της ο Όμιλος. Ε, είναι σίγουρο και το είδαμε αυτό από άλλο, από άλλο στόλο άλλης επιχείρησης ότι αυτή, αυτός, αυτή, η αλία ε, δεν είναι κερδοφόρα αλλά δεν είναι και βιώσιμη. Ε, διότι αυτή τη στιγμή διατηρείται ε, μόνο για άλλους λόγους. Σίγουρα όχι εξαιτία της τιμής στην οποία πωλείται ε, το, το ψάρι. Ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη, τα μεγάλα σούπερ συνεργαζόμαστε μαζί τους, συνεργαζόμαστε με όλο τον κλάδο. δεν πρόκειται για ρύθμιση λογαριασμών ή για... δεν σας κρύβω βέβαια ότι αυτή η μέθοδος αλίας θεωρώ ότι είναι καταστροφική και δεν το λέω μόνο εγώ. Είναι πάρα πολύ προβληματική για το περιβάλλον. Και με ανησυχεί που ε, κρατικοί πόροι χρησιμοποιούνται για να επιδοτηθεί. Είναι αλήθεια, δεν έχει γίνει κοινωνικο-οικονομική μελέτη στην Γαλλία, γιατί το θέμα δεν συζητήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Grenelle de la Mer, και γι' αυτό προσπαθήσαμε να δώσουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ε, δεν υπάρχουν, ε, δεν είναι γεμάτη λάθη, ε, ίσως υπάρχει κάποιο μικρό λαθάκι εδώ και εκεί, αλλά ο Τόνι Μπεργζέ που είναι ο λογιστής της Bloom μπορεί να μας δώσει λεπτομέρειες, μπορείτε να τον ρωτήσετε, μπορεί να σας δώσει πολλές λεπτομέρειες, είναι πρώην ελεγκτής τη Άρθουρ Άντερσεν, έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλη στερεία στη Γαλλία, στην καριέρα του μπορεί να σα απαντήσει, είναι αυτό ο οποίο ανέλησε του λογαριασμού. εγώ δεν γνωρίζω, ε, δεν είμαι λογιστής, λογιστρία. Δεν υπολογίσαμε ε, την, επιδοτήσεις κατά κεφαλήν. Αυτό δεν είναι δύσκολο όμω. Είναι εύκολο όπω λέει και ο Ντενί. Τώρα, ε, το, ο χάρτης, αυτός ο διαστρεβλωμένος ε, χάρτη. Αυτό βασίζεται στις εκφορτώσεις των βαθύβιων ειδών. Γι' αυτό το λόγο μερικές χώρες δείχνουν πολύ μικρές. Ε, κύριε Νουβιά, παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι, διότι έχουμε άλλο ένα πάνελ. Απαντάω απλώς σε ερωτήσεις. Ναι, ναι, ξέρω ότι απαντάτε, αλλά σας ζητώ να απαντήσετε πολύ σύντομα. Οι απαντήσει μπορεί να είναι πάντοτε ε, πιο μακροσκελή ή λιγότερο μακροσκελή. εντάξει. Λίγο πιο σύντομα λοιπόν. Ε, τελειώνοντας να σας πω ότι με κόβετε πάντοτε λίγο πριν τελειώσω. Τι να σας πω πρόεδρε. να σου πω ότι έχουμε το πρόβλημα όχι μόνο της μη κερδοφορίας αλλά και της μη βιωσιμότητας. Αυτό το δείχνουν τα στοιχεία μας και ελπίζω ότι θα φωτίσουν την κατάσταση. Οποιοςδήποτε μπορεί να τα δει στο ίντερνετ ε, μπορεί να δει τους ε, λογαριασμούς, ε, τους ισολογισμούς ε, και μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Πρόεδρος, ε, ναι, σα ε, σταματάω γιατί δεν τελειώνετε. Αν δεν σα είχα σταματήσει θα είχα τελειώσει. Ποιος Καντέκ. Ε, εδώ έχουμε έναν από του υπεύθυνου τη συγκεκριμένη εταιρεία και σα ζητώ, αν δέχεστε, να απαντήσει στην κυρία Νουβιό. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, μια και αναφέρθηκε η εταιρεία ονομαστικά. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε το λόγο. Σύντομα όμω. Ευχαριστώ. Η εταιρεία μας, η ΣΚΑΠΕΣ, έχει 18 σκάφη, είναι τρεις εταιρείες συνολικά. Για τον κλάδο της αλίας όσοι δεν το ξέρετε και προφανώ κάποιοι που μιλούν σήμερα δεν το ξέρουν, έχει διαφορετικέ δραστηριότητε, διαφορετικέ ζώνες, διαφορετικέ τεχνικέ, διαφορετικά είδη. Τα πιο αποδοτικά σκάφη μα είναι αυτά που εκμεταλλεύονται βαθύβια είδη. Εξ αρχή μέχρι τα, τα, ε, τα σκάφη ήταν καινούργια, μεγαλύτερα, 46 μέτρα και δίνουν 300.000 ευρώ κέρδη κάθε χρόνο. Κάθε σκάφος έχει δικό του λογιστήριο. Το, σύνολο, το σύνολο του ομίλου ΣΚΑΠΕΣ έχει θετικά ε, αποτελέσματα από το 8. Άλλες δραστηριότητες είναι λιγότερα αποδοτικές. Ξέρουμε ωστόσο ότι πολλές επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους έχουν δραστηριότητες που δεν είναι πάντα αποδοτικές. Το θέμα είναι τι γίνεται συνολικά. Ο ρόλος μας τώρα είναι να δώσουμε στον Ευρωπαίο καταναλωτή προϊόντα της θάλασσας που αλλιεύονται με βιώσιμο τρόπο, που, είναι, ε, που μπορούν να τυχνηλατηθούν και όλα τα άλλα είναι κατηγορίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόντους ζήτησε το λόγο. Κοιτάξτε, <clears throat> Έχω ενθουσιαστεί με αυτή την ακρόαση και έχω μία ερώτηση. Ε, καταρχήν προς τον κλάδο και κατά δεύτερο προς τους επιστήμονες. Αν τα κατάλαβα όλα καλά, είναι <clears throat> τραγικό το να χρησιμοποιούνται ε, τα πλάδια και οι τράτες γιατί καταστρέφεται ο βυθός. Και μία ερώτησή μου προς τον κλάδο. Τότε γιατί δεν χρησιμοποιούνται παραγάδια αφού το ξέρουν ότι αυτά είναι πολύ καλύτερα. Δεν είναι δυνατόν να καταστρέφει κανείς το βυθό για 500 χρόνια. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Και θέλω όταν βγω από αυτή την αίθουσα να έχω καταλάβει. Θα δώσουμε το λόγο στο τέλος αν έχουμε χρόνο και αν η επόμενη είναι γρήγορη. Τέταρτο πάνελ, κατευθείαν. Λυπάμαι, είστε τελευταίοι, παρακαλώ να είστε συνοπτικότατη. Ο κύριος Φράνσις Νίτ. Adelante. Παρακαλώ. Okay, thank you very much for inviting me. Um, I'll try and introduce a little bit of science back into the... Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να ε, επαναφέρω κάποια επιστημονικά στοιχεία στη συζήτηση. Εγώ προσωπικά είμαι βιολόγος αλίας ε, και δουλεύω για τη Marine Scotland ε, και για την ICES, ε, την Διεθνή Επιτροπή για την Εξερεύνηση της Θάλασσας. Και επιτρέψτε μου τώρα να σας υπενθυμίσω τις περιοχές για τις οποίες μιλάμε. Δεν αναφέραμε την ΙΑΘ που είναι η Επιτροπή του Ανατολικού Ατλαντικού. Μέσα λοιπόν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο έχουμε περιοχές ε, όπως τις νήσες, νήσους ε, Φαρόου, τα Σέτλαντ, ε, το Βισκαϊκό Κόλπο και τις Αζόρες και έχουμε το Mid-Atlantic Ridge και το Hutton Bank, την περιοχή αυτή. Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ διαφορετική ποικιλία ψαριών, πάνω από 200 είδη και το σημαντικότερο είναι ότι ορισμένα από αυτά, όχι όλα, είναι βάλωτα ε, αντικείμενο υπεραλίευσης. Στις περιοχές αυτές έχουμε λάσπη, άμμο, ε, μητρικούς βράχους, βιογενείς ε, υφάλους και εκεί ε, ορισμένες περιοχές είναι ευάλωτες, άλλες λιγότερο ευάλωτες. Κάτι που μπορούμε να πούμε για τα βαθαία ύδατα είναι ότι με το βάθος ε, μειώνεται το φως, ε, το φως μειώνεται, το ίδιο μειώνεται και η θερμοκρασία και η διαθεσιμότητα τροφής. Έτσι λοιπόν ο μεταβολισμός, η ανάπτυξη, η αναπαραγωγή, η ορίμανση, όλα αυτά καθυστερούν. Κατόπιν τούτου ε, τα ε, ψάρια αυτά είναι περισσότερο ευάλωτα. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι μας ότι έχουν υπάρξει προβλήματα ε, βιωσιμότητα σε αυτά τα είδη, γι' αυτό δεν αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Έχει υπάρξει υπερεκμετάλλευση ε, ψαριών όπως το καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού ε, και των σκυλόψαρων. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές επιπτώσεις από τα παρεπίμπτοντα αλλιεύματα και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν ή επηρέασαν κατά παρελθόν το ευάλωτο ε, οικοσύστημα, ένα άλλο οικοσύστημα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να γίνει περισσότερο βιώσιμη αυτή η αλία. Τρία βήματα. Πρώτον, ρυθμίσεις και λειτουργία της αλίας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να φτάσει σε βιώσιμα αποθέματα. Δεύτερον, προστασία των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και το τρίτον, ε, επιστημονική αξιολόγηση ε, των, ε, του περιβαλλοντικού καθεστώτος ε, και των ε, οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων. Ας δούμε το πρώτο βήμα για τους κανονισμούς και τη λειτουργία της αλίας. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό, γι' αυτό δεν θα καθυστερήσω. Πρέπει να περιστούν οι προσπάθειες και να ενισχύσουμε τα συστήματα εντοπισμού σκαφών, να απαγορεύεται η στόχευση των πλέον ευάλωτων ειδών, να απαγορευτούν οι καταστροφικές αλληλευτικές πρακτικές, να μην υπάρχουν έχουν ε, Υπάρχει κάποια πρόοδος από τότε που προέκυψε ο κανονισμός το 2003. Αυξήθηκαν οι προσπάθειες σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και βλέπουμε ότι οι αλληλευτικές προσπάθειες ε, έχουν ε, μειωθεί κατά 50%. Το κόκκινο που βλέπετε είναι οι τράτες. Επίσης, πλέον τα σκάφη δεν φέρνουν VMS και υπάρχει πλήρης απαγόρευση αλίας ε, του καθρεπτόψαρου, του Ατλαντικού και των σκυλόψαρων. Κάτι έχει γίνει λοιπόν τα τελευταία δέκα χρόνια. Το δεύτερο βήμα είναι η προστασία των ευάλωτων ενάλλειων οικοσυστημάτων. Αυτό που πρέπει να το προστατεύσουμε είναι το σύστημα αυτό, να απαγορεύσουμε τις, ε, την αλία στο βυθό, ε, σε απότομες πλαγιές, ε, και σε άλλες παρεμφερείς περιοχές. Επιπλέον, νομίζω πρέπει να προστατεύσουμε ε, και τα, ε, τους οικότοπους ε, που βρίσκονται στους βυθούς της θάλασσας. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε και τον, τις πλαγιές που ενδιαφέρουν λιγάκι από τις κοραλιογενείς περιοχές. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε σημειώσει πρόοδο στο δεύτερο βήμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ε, περιοχές ε, διατήρησης ε, με βάση το πρόγραμμα Natura 2000. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει παύσεις αλίας εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές ε, κοντά στα Βρετανικά νησιά που αφορούν αυτές τις ε, περιοχές. Έχουν, όπως σας είπα, προταθεί ή έχουν ήδη καθοριστεί ως περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η αλία δεν επιτρεπεται η αλια Bank και ε, έχουν προταθεί και άλλες περιοχές να κλείσουν. Επίσης και στον Ατλαντικό και κάποιες μικρότερες περιοχές όπως το Danway Bank στην Ισπανία. Συνολικά λοιπόν μιλάμε για 600.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από <clears throat> απαγορεύεται ελεία. Το πρόβλημα είναι ότι στην, τον Ιανουάριο ε, έχουν εκπνεύσει αυτές οι συμφωνίες και θέλω να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει μέτρα στο, να μην επιτραπεί η ελεία σε αυτές τις απαγορευμένες περιοχές. Επίσης, το δεύτερο τμήμα του δεύτερου βήματος. Εκεί προβλέπεται να προστατευτεί ο οικότοπος. Εγώ τα κρατημέλη, αλλά η Σκοτία έχει καταθέσει μία πρόταση που αφορά τουλάχιστον έξι περιοχές ε, που πρέπει να θεωρούνται ως ε, περιοχές διατήρησης της φύσης. Μεγάλες λοιπόν περιοχές που θα ισχύουν ως περιοχές διατήρησης της φύσης στο μέλλον. Το τρίτο βήμα είναι να ε, βελτιωθεί η επιστημονική βάση. Όπως βλέπετε δεν υπάρχουν αρκετά ε, στοιχεία για να βασιστούν σε αυτά οι επιστήμονες ε, ε, Πρόοδος βέβαια έχει σημειωθεί πρόσφατα και κατόπιν τούτου είναι απαραίτητο να ερευνήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ε, ενίσχυση και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εμπορικά είδη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν, ε, ακούσαμε σήμερα, πολύ καλά παραδείγματα για το πώς μπορούν να ελέγχονται κάποια είδη ε, βαθύμετρα, παραδείγματο χάρη σαν αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που συνάντησα εγώ ασχολούμενο με τα θέματα αυτά είναι η πρόσβαση σε δεδομένα ελέγχου και εντοπισμού ε, σκαφών που μας επιτρέπουν να έχουμε το αποτύπωμα των σκαφών. Σήμερα ε, δεν υπάρχει καλή πρόσβαση σε αυτό και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Όσον ε, αφορά τα ψάρια, ακούσαμε πάρα πολλά από το πρόγραμμα Deep Fishman που έχει ως στόχο να βελτιώσει την κατάσταση για κάποια είδη. Η Σκοτία δεν έχει κάποια ανεξάρτητη μελέτη. Ε, βέβαια, ε, σε κάποια αποθέματα παρουσιάζεται μείωση, σε άλλα πάλι αύξηση. Ε, βλέπετε εδώ τα παραδείγματα ε, όπου διαπιστώσαμε σημαντική αύξηση αποθεμάτων τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που βλέπετε είναι ο καρχαρίας της Πορτογαλίας, είναι ένα πολύ ευάλωτο είδος και δεν βλέπουμε εκεί να έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην επάρκεια αυτού του είδους, στην πυκνότητα αυτού του είδους. <clears throat> Ας δούμε τους ε, οικότοπους. Έχουν ε, κλείσει μεγάλες περιοχές και οι τελευταίες ε, μελέτες, ο κύριος Ρίβερ μίλησε επ' αυτών, έδειξαν ότι υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα για τα ευάλωτα ενάλια οικοσυστήματα. Αυτό που βλέπετε είναι το North Work, Work Closure, Αυτό συγκεκριμένα είναι 30 χιλιόμετρων. Ε, δεν έχουμε στοιχεία ε, βαθύμετρου, από το βαθύμετρο και δεν ξέρω, εδώ μπορείτε να δείτε ένα βίντεο σχετικά με το αποτύπωμα που έχουμε στα χέρια μας. Μιλάμε για έναν κορεαλιογενή υφαλό 70 μέτρων με πολύ ειδικέ συνθήκες. Το αποτύπωμα του κυρίου River είναι πολύ καλύτερο βέβαια από το δικό μας μπορούμε να διαιτηθούμε κατά πόσον αρκούν όλα αυτά έτσι ώστε ε, οι πράξεις μας να είναι οικολογικά βιώσιμες. Ε, θεωρώ ότι ε, θα υπάρχει σύντομα πολύ μεγάλη προστασία. Υπάρχουν κάποια βατήδια είδη που παρουσιάζουν κάποια βιωσιμότητα, όμως τα πλέον ευάλωτα ήδη ακόμα και των σταθερών είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα όπως σας είπα το καθρεπτό ψάρο του Ατλαντικού και τα σκυλόψαρα. Ε, γι' αυτά πρέπει να υπάρξουν ειδικά μέτρα προστασίας και εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα των απορρίψεων. Έχουμε εργαστεί με το θέμα αυτό και έχουμε διαπιστώσει ότι η βιοπικιλότητα, η ποικιλία τους φτάνει μέχρι τα 1.500 μέτρα. Έτσι λοιπόν ε, οι απορρίψει είναι πολύ ψηλέ σε αυτά τα επίπεδα. Τι θα κάνουμε τώρα στο μέλλον. Ε, προσπάθησα ε, να δω τι σημαίνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως η Αλία με τις τράτες. Θα επιτρέπεται η χρήση σε κάποιες συγκεκριμένες τράτες, σε κάποια συγκεκριμένα είδη για, το, ε, βραχό, για, το, για την πεσκαντρίτσα, αλλά για το γρεναδιέρο θα επιτρέπετε μόνο το 10% να λιεύεται. Αυτό που θα επιτύχει η πρόταση είναι ε, να υπάρχουν πολύ λίγα κίνητρα ε, για τις στράτες ε, στα, που ασχολούνται με την αλληλεία βαθέων υδάτων. Τώρα, πώς μπορεί να υπάρξει ανασύσταση. Νομίζω ότι τα ευάλωτα είδη καλύπτονται καλύτερα εφόσον υπάρχει απαγόρευση αλίας. Υπάρχουν τα, οι κορολογενείς υφαλή που σας έδειξα προηγουμένως. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση αυτή ε, θα είναι ιδιαίτερα ε, επικερδής και υποφελής ε, για τα ευάλωτα είδη. Όμως θα επιτρέψει τη μείωση των απορρίψεων ευάλωτων ειδών, γιατί σας είπα κυρίως ότι αυτά εμφανίζονται στα 1000 με 1500 μέτρα. Δεν θα υπάρχουν κίνητρα για την αλία σε αυτό το βάθος. μπορούμε να δούμε εναλλακτικέ τεχνικές αλίας. Αυτές αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν πιστεύω ότι τα παραγάδια είναι καλύτερα γιατί αυτά ε, κόβουν, ε, τα πληγώνουν και κατακρεοργούν τα, ε, τους καρχαρίες. Ίσως μπορεί να γίνει κάποια προσαρμογή για το θέμα αυτό. Θα ήθελα τώρα να δούμε λιγάκι τις εναλλακτικές λύσεις ένα από τα προβλήματα που έχω διαπιστώσει με την πρόταση αυτή είναι ότι ε, το παράδειγμα 1 ε, περιλαμβάνει ήδη ε, που μπορούν να την χάνουν αλίες και βιώσιμης αλίες, όπως η μουρούνα. Αυτό που έχει σημασία είναι να περιορίσουμε την αλία το ανώτερο μέχρι τα χίλια μέτρα. Και σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ. Το βλέπετε αυτό, το έχω πει ε, και σε όλες τις γλώσσες ε, που μπορούσα να το πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζιάννη, τελευταίος ομιλητής. Παρακαλώ και αυτός όσο περισσότερο ε, συνοπτικός είναι. Και ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω. Να πω πριν δώσω το λόγο. Ζήτησα λίγο περισσότερο χρόνο από τους διερμηνείς που μας δίνουν 10 λεπτά ακόμα για να τελειώσουμε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω στα αγγλικά. Είμαι σύμβουλος της Συμμαχίας για τη διατήρηση του Deep Sea Conservation. Έχουμε πολλά μέλη, κάποια τα βλέπετε, τα ξέρετε. Επίσης είμαι και consultant στον ε, ΦΑΟ του ΟΗΕ το IUCN και έχω, έχω δημοσιεύσει μια σειρά εκθέσεων σχετικά και έχω συμμετάσχει σε μια σειρά διεθνή, διεθνών ε, διασκέψεων. Δύο φορές έχω έρθει στην Επιτροπή σας στο παρελθόν για παρουσιάσει στο θέμα αυτό, το 4 και το 7. Χαίρομαι που έχω τη χαρά να είμαι ξανά εδώ. Ήμουνα εμπορικός ψαράς για 7 χρόνια, 5 από τα οποία σε βαθιά νερά. Τα τελευταία 10 χρόνια έγιναν αρκετέ διαπραγματεύσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ για το θέμα αυτό, εκτεταμένε. Πολλέ φορέ το εξέτασε η Γενική Συνέλευση το θέμα αυτό. Και το θέμα που εξέτασε ήταν η βιωσιμότητα τη αλληλεία, η προστασία τη βιοποικιλότητα, η δικαιοσύνη και η εφαρμογή τη διεθνή νομοθεσία. Θέματα δηλαδή που εμπολί συζητούνται και εδώ σήμερα. Παρόμοιε ήταν και οι ανησυχίε με αυτέ που τέθηκαν από άλλου ομιλητέ. Δεν θα τους, ε, δεν τι αναφέρω, αλλά να πω απλά ότι εμπολεί τα βαθύ, η βαθύ βιαλή είναι διαφορετική από την παράκτια, την πελαγική και την υπηρετική αλληλεία τόσο για τη διαχείριση της αλίας και για τον αντίκτυπο της αλίας στα οικοσυστήματα. Μετά από 10 χρόνια συζητήσεις στον ΟΗΕ, πρόκειψαν τέσσερα ψηφίσματα. Και άλλα είναι, αλλά τα τέσσερα είναι τα βασικά. Η συζήτηση συνεχίζεται προφανώ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η βασική συμφωνία έλεγε να αποφευθεί σημαντικές αντίξωες επιπτώσεις ευάλωτα ενάλια οικοσυστήματα με περιβαλλοντική ε, με μελέτη αντικτύπου πριν γίνουν, ε, ξεκινήσει η αλληλεία, τη δημιουργία περιοχών κλεισί, προληπτικού κλεισίματος όπου υπάρχει κίνδυνος ε, ευάλωτων περιοχών και να κλείσει η περιοχή μέχρι να υπάρξουν μέτρα, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αλληλευτικών αποθεμάτων βαθέως θαλάσσιας συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένα είδη, και τον κανόνα του Μουβών. Η Γενική Συνελεύση ήταν σαφή. Ε, και όταν λέω Γενική Συνελεύση, λέω Γενική Συνελεύση δηλαδή τα κρατη έτσι, το άθεσμα των κρατών Τα, τα ψηφίσματα αυτά υιοθετήθηκαν μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ ε, κρατών που έχουν αλία, ε, βαθύ βιαλία και κρατών που έχουν εκτεταμένα, εκτεταμένες ακτές και η Ένωση συμμετείχε δραστήρια σε όλα αυτά. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και πάλι, αλλά μπορώ να σας πω τα μέτρα που συμφωνήθηκαν από την συλλογική διεθνή κοινότητα στον ΟΗΕ βασίζονται σε κάποιες βασικές ε, ρυθμίσεις της σύμβασης για το, για το νόμο, της, ε, το, για το νόμο περί διατήρηση, διατήρηση του, και προστασία του περιβάλλοντος, αποφυγή δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις στο ενάλλειο περιβάλλον. Η συμφωνία επίσης στηρίζονται σε κάποιες βασικές ε, ρυθμίσεις της συμφωνίας για τα, αλλιεύματα, για τα ε, αποθέματα αλλιές του ΟΗΕ, για την ε, ρύθμιση της Ελίας και στο ανοιχτό και στα διεθνή ύδατα και στην ε, ε, αποκλειστική οικονομική ζώνη με προστασία ε, της βιοπικιλότητας, βιώσιμη διατήρηση των αποθεμάτων, εφαρμογή της αρχής της πρόληψης, προστασίας της, ε, των οικοσυστημάτων κλπ. Βασικό είναι το τελευταίο που έβλεπε τη σελίδα αυτή. Η απουσία επαρκούς ε, ενημέρωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως, ρόζος, ως λόγος αναβολή, αναβολής ή μη λήψης μέτρων διατήρησης ή διαχείρισης. Κάτι που η Ένωση υιοθέτησε το 2003. Το άρθρο 7 της συμφωνίας αυτής επιπλέον μιλά για την ε, υιοθέτηση συμβατών μέτρων και στα διεθνή ύδατα και στα χωρικά ύδατα, τονίζοντας ωστόσο εδώ ότι τα περισσότερα αποθέματα, βαθύρια αποτέλεσμα, από, αποθέματα, ε, ε, αντλούνται από το βορειοανατολικό Ατλαντικό πέραν ε, της Γενικής Συνέλευσης των ΟΗΕ είχαν και μια, και μια παράλληλη διαπραγμάτευση υπό την ε, αιγίδα του ΦΑΟ. Το 2006 όταν η Γενική Συνέλευση συμφώνησε μεταξύ των παράκτιων χωρών και των λευτικών χωρών ότι η διαλύεια θα πρέπει να την χάνει διαχείριση για να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο ενάλλειο περιβάλλον μέσω ε, της διεξαγωγής ε, με ε, αξιολόγηση αντικτύπου. Το βασικό ερώτημα ήταν πώς γίνονται οι μελέτες αντικτύπου, πώς εντοπίζουμε τα ευάλωτα οικοσυστήματα. Οπότε κάτω από το ΦΑΟ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις όπου και πάλι μετήχαν όλα τα παράκτια, όλα τα ε, βαθύ, τα, τα κράτη με βαθύ βιαλία και κάποια παράκτια κράτη που έδωσε διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τη, για τη βαθύ βιαλία. Τα guidelines που λέμε. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα εργαλείο διακυβερνητικό και όχι ε, συνθήκη. Είναι μια, ένα αποτέλεσμα μακρών διαπραγματεύσεων. Εδώ περιλαμβάνονται κριτήρια για μελέτη αντικτύπου, για τον καθορισμό των ε, ε οικοσυστημάτων που κινδυνεύουν. Το 9 ή το ψήφισμα 64-72 του και 72 της Γενικής ζητούσε να ληφθούν μέτρα βάσει των καθηγητήρων των γραμμών. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αυτά είναι τα κριτήρια ωστόσο για τον, τη μελέτη αντικτύπου. Η συμφωνία υπογράμμιζε δηλαδή ότι αυτέ οι μελέτε αντικτύπου πρέπει να, πρέπει να γίνονται πριν ξεκινήσουν ε, οι δραστηριότητε αλεία, ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα πριν δοθούν οι άδειε. Χάνω κάποιε σελίδε πέραν ωστόσο του τι γίνεται σε διεθνέ επίπεδο. Κάποιοι κανονισμοί τη Ένωση άρχισαν να εφαρμόζονται, να υλοποιούνται. Ο 237 του 2002, για το καθεστώς πρόσβαση στα βαθύβια ύδατα, ο 156 που απαγόρευσε την, ε, τα απλά διαβυθού και ειδικά εργαλεία για τη Μαδέρα και τις Αζόρες. Ο 732 του 2008 που εφαρμόζει το ψήφισμα του ΙΕ 105 για περιοχές των των διεθνών υδάτων όπου επιτρέπεται η αλλιεύση χωρίς περιφερειακή οργάνωση διαχείριση αλλιές για την αντιμετώπιση και διαχείριση τέτοιας μορφής αλλιές και ο 43 του 2009 κανονισμός του Συμβουλίου που επιτρέπει, που απαγορεύει την, ε, ε, τα απλάδια, σε, το ψάρεμα με απλάδια κάτω των 600 μέτρων. Μπορείτε να δείτε όλα αυτά τα στοιχεία και στην ιστοσελίδα μας. Απλά εγώ σας δίνω κάποια στοιχεία από τη UNEP και από εμά για τη, τις επιπτώσεις της ε, αλίας. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κάθε μορφή αλίας έχει αντίκτυπο στον πυθμένα των α, θαλασσών, αλλά βέβαια τα απλάδια είναι τα, το, τα πιο επικίνδυνα. το ISIS το έφερε, το αυτό το θέμα τα τελευταία 10 χρόνια όντω. Εδώ είχατε μία φωτογραφία, μία σειρά φωτογραφιών, θα είχατε μία σειρά φωτογραφιών από τα ενάλληλα συστήματα, αλλά δεν τα βλέπετε. Φωτογραφίες ήταν πάντως ε, αρχαίγωνων κορεγινών περιοχών που άλλαξαν μετά οι Νορβηγοί το πήραν αυτό και μην τονίσετε ότι οι Νορβηγοί έκτιμα ότι ήδη έχουν χάσει 30 με 50% των κοραγιών της από αυτή τη μορφή αλίας. Άλλο θέμα που εμφανίστηκε και από άλλη οπτική γωνία είναι τα παρεπόμενα διεύματα. Οι πίνακες αυτοί έρχονται από μία μελέτη ε, που ανέφερε ο κ. Βίβερ. Έρευνε σε μία περιοχή της ε, ε, Ιρλανδικής θάλασσας, στην περιοχή Porcupine, πριν και δέκα χρόνια μετά την βαθύβια αλία. 77 ήδη βρήκανε, τον οποίον η ακτίνα βυθού ταυτιζόταν με την ακτίνα ε, της ε, αλίευσης με απλάδια, μέχρι 1500 μέτρα δηλαδή, από 500 μέχρι 1500. Η μείωση κατά μέσο όρο ήταν 69%. αλλά από τα 77 ήδη 14 μόνο αντιμετωπίζονται από τον κανονισμό του Συμβουλίου. Για τα υπόλοιπα δεν υπάρχει καμία ρύθμιση και το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα ίδια αυτά. Αν η υποχρέωση για, τη διαχείριση, για τους διαχειριστές και τους νομοθέτες είναι να εξασφαλίσουν ότι, ότι προστατεύονται και τα εμπορικά και τα παρεπόμενα ρεύματα, πρέπει την απόκληση αυτή να την αντιμετωπίσουμε. Και η ISS έλεγε πάντα ότι μέχρι πρόσφατο το 100% των ε, παρεπιπτών των αλλιευμάτων ήταν εκτός ε, του ορίου ασφαλών βιολογικών, του, των ασφαλών βιολογικών ορίων. Και πάλι, ρωτάω, τι γίνεται με τα άλλα 77 είδη. συνοπτικά, κλείνοντας. Πέραν της νομικής διάστασης, υπάρχει και ενδιαφέρον από πλευράς της κοινή γνώμης αρκετά χρόνια. Υπήρχε μια ε, συλλογή υπογραφών ΑΒΑΖ, 705.000 ε, υπογραφές ε, για την απαγόρευση της βαθύβιας βιασαλίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός υπογραφών που μάρεψε αυτή η οργάνωση ΑΒΑΖ, κυρίως από κράτη μέλη της Ένωσης. Υπήρξαν σειρά δηλώσεων επιστημόνων που ζήτησαν κάτι αντίστοιχο, ένα μορατόριο βασικά, 130.000 υπογραφέ. Κάποιε κάποιες ε, σούπερ μάρκετ άραξαν την πολιτική αγορά ε, και ο Μπράνσον ακόμα είχε στείλει ένα γράμμα στον Υπουργό Μπένιον. Ε, υπήρχε μια δήλωση των εμπλεκομένων φορέων με πάνω από 500 υπογραφίε, περισσότερε από όσε βάδα μαζέψαμε εμεί δηλαδή, πριν έρθουμε εδώ. Και τα μέσα ενημέρωση έδειξαν ενδιαφέρον και τέλο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕΦ επανέλθει στο θέμα το 2015. Η χρονική στιγμή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή γιατί και η δική σας ε, συζήτηση περίπου τότε θα τελειώσει. Φαντάζεστε ότι έχω μια σειρά συστάσεων που τηρούν ε, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που ζητούν να υπάρχουν ε, αξιολόγηση αντικτύπου για όλα τα, για όλα τα να, να υπάρχουν περισσότερες ε, δυνατότητες ε, αλληλευτικής, δυνατότητες όπου υπάρχουν, να μην υπάρχουν αλληλευτικές δυνατότητες να υπάρχουν στοιχεία, μέτρα για, την, για τη μείωση των παρεπόμενων αλληλευμάτων κτλ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Για το θέμα του ορισμού εμείς προτείνουμε το, τα 200 μέτρα. Ευχαριστώ πολύ που τρέξατε. Δύο-τρία λεπτά έχουμε ακόμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Αρσένη έτσι ώστε σε ένα λεπτό να κλείσει για να τελειώσουμε. Έχουμε ξεπεράσει το ωράριό μας. Έτσι κι αλλιώς ο 8 συν 3 ομιλητέ, 25 ε, ε, ευρωβουλευτέ που μίλησαν, οι απαντήσει των ομιλητών, πώς θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Κύριε Αρσένη, ε, ζητούμε και συγγνώμη για αυτούς που είχαν ερωτήσει και δεν πρόλαβαν να τι θέσουν. Ελπίζω όλοι όμως να ρώτησαν αυτό που ήθελαν να ρωτήσουν και να πήραν την απάντηση. Ο στόχος ε, της ακρόασης νομίζω ότι επετεύχθη ε, μέχρι το τέλος η συμμετοχή ήταν ζωντανή ε, η βιωσιμότητα, μακρόχρονη βιωσιμότητα των βαθύβιων ειδών είναι ο στόχος μας. Είναι σαφές ότι η πρόταση που έχουμε ε, οδηγεί σε αλλαγή των αλληλευτικών εργαλείων προκειμένου να αποφύγουμε απαγόρευση μιλούμε για αλλαγή εργαλείων έτσι ώστε να συνεχίσουμε να αλλιεύουμε χωρίς αρνητικές ε, επιπτώσεις. Και μιλούμε για ε, αλλαγή εργαλείων ε, προς εργαλεία που βοηθούν, που είναι πιο πολύ βιώσιμα οικονομικά, αλλά βοηθούν και στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Παράδειγμα για παραγάδια. Εθίχησαν πολλά πράγματα, πολλές ερωτήσεις, πολλά ερωτηματικά. Ε, καταλαβαίνω πολύ καλύτερα πια το, το θέμα των ποσοστώσεων ή ποσοστώσεις δεν έχουν άμεση σχέση με το πράγμα τη Κομισιόν. Διαπιστώσαμε πόσο μεγάλο είναι πόσο σημαντικές είναι οι συνέπειες ε, είδαμε τις διαφορές ανάμεσα σε τράτες και παραγαδιά. Ε, νομίζω η ήταν πολύ πλήρης, ε, πολύ τροφή για σκέψη, προκειμένου να απαντήσουμε αποτελεσματικά και συγκεκριμένα ως Κοινοβουλίο. Ευχαριστούμε κύριε Αρσένη, λέει ο Πρόεδρος. 30 δευτερόλεπτα. Η κυρία Λεβέν ήθελε να θέσει ένα θέμα, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας, να σας ζητήσω να αναβάλουμε την προθεσμία για τροπολογίες για τον κανονισμό για τα χέλια, δεδομένου ότι ε, στην στη συνάντηση Επιτροπής ε, ε, ακούστηκαν διάφοροι δισταγμοί, κάποιες επιφυλάξεις. Η, η, προθεσμία έλγε τη Δευτέρα. Θα ζητούσα περισσότερο χρόνο για να έρθω σε επαφή με τους και πριν τη λήξη της προθεσμίας. Συνεπώς θα μπορούσαμε να αναβάλουμε αυτή την προθεσμία, αυτή τη λήξη. Δεν χρειαζόμαστε μία εβδομάδα, χρειαζόμαστε ένα μήνα τουλάχιστον. Υπάρχει καμία αντίρρηση γι' αυτό? Όχι. Ωραία. Σύμφωνοι. Θα το, θα το... θα ενημερώσουμε δημοσίως για τις, ε, αποφασίσεις των συντονιστών, για τις των συντονιστών τις έχετε πάρει, δεν υπάρχουν θέματα, θεωρούνται εγκεκριμένες. Επόμενη συνάντησή μας 20 Μαρτίου το πρωί και το απόγευμα και 21 Μαρτίου μόνο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα στους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.